λαμβανθούν υπόψη τα πρότυπα ε, τα αναπτυξιακά για τη νέα διεθνή διακυβέρνηση. Θα ακούσουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των βασικών συστάσεων αυτής της μελέτης και στη συνέχεια τα σχόλια της Επιτροπής και του Concord πριν να ξεκινήσει η συζήτηση ανάμεσα στους ε, βουλευτές. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Πέντρο Μορασάν. Παρακαλώ έχετε 10 λεπτά Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η μελέτη που θα σας παρουσιάσω συνοπτικά εκπονήθηκε από δύο φορείς της ΕΠΣ των Βρυξελών, Σούτβιν και είμαστε παρόντες οι τρεις συντάκτες έκθεση, ο κύριος Πέρενς, η κυρία Φρεντερίκ Νίβερτ και ο υποφαινόμενος Πέδρο Μορασάν. Εμείς καταρτήσαμε την έκθεση, οπότε είμαστε και τρεις στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε απορίες σας. Πολύ συνοπτικά λοιπόν, γιατί ένα δεκάλεπτο είναι ανεπαρκές για να καλύψει την περιπλοκότητα αυτής της έκθεσης. Θα προσπαθήσω πάντως να κάνω μια ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων και των συστάσεων που έχουμε να υποβάλουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το όλο πλαίσιο, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, και επίκαιρο, γιατί ο καθορισμός ενός νέου θεματολογίου μετά το 2015 θα ήταν πρόκληση για τον επαναπροσδιορισμό της επίσημης ε, βοήθειας για την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα όταν ζητούμενο είναι να γίνει μια λειτουργικοποίηση της ιδέας της διεθνούς κοινότητας για κοινέ αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες δυνάμει των ικανοτήτων των δωρητών, που είναι πολύ και διάφοροι, αλλά και των χωρών εταίρων που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Από την άλλη πλευρά, το όλο κλίμα και το τοπίο της διεθνούς συνεργασίας και η κατάσταση της διεθνούς συνεργασίας έχει αλλάξει άρδιν εμφανίστηκαν νέοι φορείς, νέοι παράγοντες, ε, νέα εργαλεία, καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και οι αναδυόμενες οικονομίες άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερο δωρητές. Έτσι τροποποιήθηκαν τα ποσοστά συνεισφορά στην παγκόσμια και βοήθεια. Επίσης ε, η κινητοποίηση εχώριων πόρων των ε, χωρών εταίρων και δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων έχουν ε, αναγνωριστεί ως, τη βασικ... ως η βασικότερη πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Κάτι που αυτόματα μειώνει τη σημασία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, της ΩΝΤΑ. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά της, αναπτυξιακ... της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη εμ, καθιστούν παροχημένη ε, την έννοια αυτή τη όντα που είχε διαμορφωθεί το 1969, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο που έχει λάβει τώρα η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, ο ισχύων ορισμό τη όντα, της επίσημης αναπτυξιακή βοήθειας, καλύπτει και τη στρατιωτική βοήθεια υπό όρους, κάποιες αντιτρομοκρατικέ δραστηριότητες, ειρηνευτικές αποστολές, πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, καθώς και πολιτιστικά προγράμματα και υποτροφίες αν ακολουθούσαμε στελτική ερμηνεία του ορισμού της επίσημης αναπτυξιακής βοηθείας, όλα αυτά τα πεδία θα καλύπτονταν. Αυτό βέβαια μπορεί να επιδέχεται διπλή ερμηνεία με τον νέο ορισμό. Γι' αυτό και η πιο έντονη κριτική σχετίζεται με τα θέματα της κοινή δωρεάς για την αναδιάρθρωση του χρέους, το κόστος για τους πρόσφυγες, γιατί είναι θέσεις που καλύπτονται από την αναπτυξιακή βοήθεια, αυτή την επίσημη, επίσης ανθρωπιστική βοήθεια, τεχνική συνεργασία και αρρωγή. Όλες αυτές οι κριτικές ε, δεν μπορούν να αγνοηθούν γιατί μερικές φορές είναι δικαιολογημένες και εύλογες αυτές οι κριτικές και προέρχονται όχι μόνο από την κοινωνία των πολιτών αλλά και από πανεπιστημιακούς κύκλους. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το επιχείρημα ότι μερικές φορέ γίνεται κατάχρηση του εθελοντικού χαρακτήρα του είδους των πληροφοριών που θέτουν οι δωρητές ε, στην αρμόδια επιτροπή του ΟΣΕ, και ΚΑΤ, της Επιτροπή της Επιτήσιας Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας, αλλά ο ισχύων ορισμός δεν αρκεί ούτε για να λάβει υπόψη τους νέους, ε, το νέα διάσταση, τις νέες διαστάσεις, αλλά ούτε και για να καταμετρήσει την αποτελεσματικότητα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Μερικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι το ισχύον περιεχόμενο της όντα μερικές φορές ε, δεν ε, αντικατοπτρίζει σωστά ή μερικές φορές ε, δεν ε, καλύπτει ούτε με ακρίβεια όλες τις πτυχές. Και μάλιστα σε μερικές φορές κάποιες έννοιες για τα δάνεια που παραέχονται στηρίζονται σε παλιούς ορισμούς και μάλιστα σε επιτόκια 14-15%, επιτόκια του παρελθόντος που δεν έχουν καμία σχέση με την παρούσα κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και μια και οι βάση του υπολογισμού των ε, δανείων αυτών ε, βαρύνει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, οι περισσότεροι δωρητές ε, αντιμετωπίζουν αυτή την έλλειψη αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε και τον αντίστοιχο ηθικό κίνδυνο. Επίσης, η ΟΑΣΕ προσπάθησε να... Η ΟΣΑ μάλλον προσπάθησε να τροποποιήσει τον ορισμό προσθέτοντας την ειδική βοήθεια χώρα προκειμένου να φέρει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια πιο κοντά στην ουσία της, που είναι η μεταφορά πόρων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η πρόοδος θα πρέπει να τύχει αναγνώριση και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις του, της έννοιας της βοήθειας, γιατί η ανάγκη της μεταρρύθμισης έχει αναγνωριστεί και από την κοινωνία των πολιτών και από τους εμπειρογνώμονες, αλλά και από την ίδια Επιτροπή ε, του ΟΣΑ, αλλά και τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία μελέτη της CCDPM μετά από εντολή της ε, Ολλανδικής και της Γερμανικής κυβέρνησης ε, αναλύονται οι αδυναμίες της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και προτείνονται δύο εναλλακτικέ λύσεις ενδιαφέρουσες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πρώτη είναι η πιθανότητα να θεσπιστεί ένας ε, γενικός δείκτης που καλύπτει την όντα με, την με τον ισχύοντα ορισμό, αλλά και τρεις άλλες μορφές σημαντικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, που περιλαμβάνουν ε, τα ιδιωτικά κονδύλια συνδρομής, επίσημα, τα επίσημα κονδύλια που δεν αφορούν δάνεια και ιδιωτικά που δεν αφορούν δάνεια, ε, που θα ελάμβαναν το χαρακτηρισμό της εξωτερικής ε, αρρωγής για την ανάπτυξη και ενισχύουν τη διαφάνεια. Οπότε κρατάει το ρισχεντορισμό της όντα, αλλά διευρύνει κάπως το, το πεδίο. Η δεύτερη εναλλακτική λύση που προτείνει η έκθεση της ACDPM είναι πιο φιλόδοξη, γιατί απαιτεί ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση του ορισμού, του ισχύοντα ορισμού της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Με βάση την ε, λύση αυτή θα πρέπει ο ορισμός να είναι πιο ανοιχτός, ώστε να περιληφθεί και η χρηματοδότηση για τις κλιματικές αλλαγές, ε, το κόστος εξασφάλισης της ιδιωτικής χρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Η Concord με ευρύτατη ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θεωρεί σε αντίθεση με την έκθεση της ACDPM να αποκλείσουμε τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης από τον ορισμό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για να, για να υπερτονιστεί ως συμπληρωματικό και έκτακτος χαρακτήρας αυτού του είδους χρηματοδότηση όπως είχε συμφωνηθεί στα πλαίσια του Μοντερέι και της Δόχα. Έχουμε και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προσανατολίζεται σε ένα συνεπές ε, σύστημα πληροφοριών για τη χρηματοδότηση, για την ε, κρίζωση της φτώχειας και την αηφόρο ανάπτυξη. Είναι πάνω απ' όλα σημαντική έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει στην ανακοίνωσή της να, να τονιστεί ο χαρακτήρας μεταφοράς κονδυλίων που έχει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το χαρακτήρα μεταφοράς των κονδύλιων της όντα. Δεύτερον, να τηρηθούν, να τα ε, κριτήρια του Μοντερέι για τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης και τρίτον, να συμβάλλουμε σε, μια, σε ένα νέο χαρακτηρισμό της παραχώρησης και επίσης να δώσουμε εξέχοντα και, εξέχουσα και περίοπτη θέση στη χρηματοδότηση του περιβάλλοντος. Η στάση μας είναι η εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δημιουργηθεί ένα αηφόρο και βιώσιμο πλαίσιο, ώστε να, τονιστεί ο χαρακτήρας της μεταφοράς των κονδυλίων του, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ώστε να ληφθεί υπόψη και είναι του CPA που έχει αναπτύξει όσα. Δεύτερη σύσταση, να συμβάλλεται στην αναθεώρηση του καταλόγου των χωρών αποδεκτών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ώστε ο στόχος ε, της ε, φόρου ανάπτυξης και της εκρίζωσης της φτώχειας να περιοριστεί στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της φήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρώντας ε, τις υποσχέσεις της διάσκεψης του Μοντερέη δηλαδή κρατώντας ε, τον συμπληρωματικό και προσθετικό χαρακτήρα των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης. Τέταρτο, θα πρέπει να επιμείνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε ο, η υιοθέτηση του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να συμβάλλει στην ενίσχυση του αντικτύπου και της προσθέμενης αξίας του όντα χωρίς να επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Πέντε, να καθοριστούν σαφέστατα τα όρια μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνει έκκληση για ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση του ορισμού της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας χάρη μιας στρατηγικής αηφόρου ανάπτυξης και όχι απλώς για να βελτιωθεί η εικόνα των δωρητών είτε είναι αυτή ε, δημόσιοι ιδιωτικοί φορείς. Επίση, μια διαφοροποιημένη διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι εξή πτυχέ. Καταρχήν, ευθυγράμμιση με το νέο θυματολόγιο για μετά το 2015. Δεύτερον, ευθυγράμμιση με τι προδιαγραφέ τη EATI και τη ε, Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη. Τρίτον, ε, θέσπιση κριτηρίων ε, πληροφόρηση για να εντοπιστεί η φύση των, των καινοτόμων πηγών και ενίσχυση του ρόλου του CPA. Επίσης θα πρέπει να στηρίξει τη θέσπιση ενός ανεξάρτητου παγκόσμιου φορέα που θα είναι διαφανής και θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες. Έβδομο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει το διάλογο με τις ε, με τους νέους δωρητές, ώστε να δημιουργηθούν ε, συνενετικές λύσεις που θα εξυπηρετούν τις χώρες αποδέκτης επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και επίσης ε, για να είναι ευρεία και σημαντική η συμβολή θα πρέπει στην αναθεώρηση του προγράμματος του 2015 να ληφθούν υπόψη τα δύο κεντρικά έγγραφα για την ανάπτυξη που είναι το θεματολόγιο για την μεταρρύθμιση και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που μέχρι στιγμής ε, δεν προσανατολίζουν, δεν συνδέουν ε, το πρόγραμμα, το στόχο της εκρίζωσης της φτώχειας με το στόχο της εφόρου ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της... Δεν ακούγεται η Πρόεδρος. Έχετε πέντε λεπτά. Δίνει το λόγο στον επόμενο μιλητή. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Πρόεδρε, ε, λέγοντας ότι για μας είναι πολύ κέρια αυτή η μελέτη. Φτάνει σε μια στιγμή όπου ξεκινάμε σοβαρές και σημαντικές διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβανομένων βέβαια των διαπραγματεύσεων για την επόμενη διαπραγμάτευση για το μελλοντικό ACA αλλά και τις μελλοντικές συζητήσεις για την εξέλιξη στο πλαίσιο των συζητήσεων μετά το 2015 στην Νέα Υόρκη. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες αν και ξεχωριστές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, της, το σενάριο νέων εξελίξεων όπως λέγεται και στην μελέτη όπου προβλέπεται η απομάκρυνση από την παραδοσιακή προσέγγιση βορρά-νότου που βασίζεται στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και να λάβουμε υπόψη ότι δεν μιλάμε πλέον για ανάπτυξη αλλά για βιώσιμη ανάπτυξη δεν εστιάζουμε πια μόνο στο input αλλά και στα επιδόσεις, στα αποτελέσματα και ότι δεν μιλούμε πλέον μόνο για επιδοτήσεις και οικονομικές και χρηματοπιστωτικές μεταφορές, αλλά και για νέα μέσα πιο περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο έχω να, κάνω, να, να, να δώσω τέσσερα σημαντικά μηνύματα. Το ένα είναι αυτό που μόλις είπα, ότι νέο χρηματοδοτικό σύστημα και νέος ορισμός της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλα αυτές τις, όλα αυτές τις διαφορές και την πραγματικότητα. Δεύτερον, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να είναι καθολικό, συνολικό, ε, να περιλαμβάνει όλες τις ροές, όχι μόνο την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και άλλες βοήθειες όπως η ροή νότου-νότου. Θα πρέπει να εξαλείψουμε οποιαδήποτε ε, ε, οποιασδήποτε παραμέτρους αλλοιώνουν τα πράγματα και βεβαίως να, όπως για παράδειγμα τις εγγύσεις και βέβαια να βελτιώσουμε την διαφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να μπούμε σωστά στις διαπραγματεύσεις. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι τομείς στην μελέτη αυτή που θα ήθελα κάποια μεγαλύτερη σαφήνεια γιατί πιστεύω πως επικρατεί κάποιες φορές σύγχυση στη μελέτη αυτή ανάμεσα στην έννοια της, του, του, του ODA δηλαδή της επίσημης αναπτυξικής ροής που είναι μια μέτρηση κάποιων ροών, τις δεσμεύσεις τις, που κάποιοι δωρητές δηλαδή ανέλαβαν φτάνοντας το 0,7% η Ένωση για παράδειγμα, καθώς και τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση για τη σχετικά, σχετικά προγράμματα, πολύ ευρύτερο αυτό από ότι απλά η επίσημη το βοήθεια και κάποιες φορές τα χρησιμοποιούνται αδιακρίτως αυτά στη μελέτη. Κάτι ακόμα που είναι πολύ τεχνικό και δεν θα μπω μέσα στις λεπτομέρειες είναι ότι Πιστεύουμε πως υπάρχουν μερικές ανακρίβειες στη συζήτηση για τις εκχωρήσεις. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή για την Ένωση. Πολύ σημαντικό να δεχτούν οι Ευρωπαϊκοί, ο ΣΑ μάλλον, τις ε, επενδυτικούς κανόνες της Ένωσης. Με κάποια επιτυχία το κάναμε αυτό, Οπότε υπάρχει ένα ε, ποσοστό ενισχύσεων, όμως κατά τη γνώμη μας αυτό που αναφέρεται στην έκθεση δεν είναι 100% ακριβές. Τώρα, για σε πολιτικές συστάσεις, συστάσεις μάλλον επί των πολιτικών, να πω ότι τα βασικά μου σχόλια ε, είναι ε, ότι θα πρέπει να τονίσουμε τα ωφέλη για την χώρα αποδέκτη, ναι, αυτό συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν και οι προσπάθειες για παρακολούθηση των δωρητών. Και τα δύο δηλαδή θα πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν επίσης κάποιες κατηγορίες χωρών για τις οποίες επίσημη αναπτυξική βοήθεια είναι πιο σημαντική και άρα ε, θα πρέπει να τονιστούν περισσότερο όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η οι ευάλωτες. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση των ενισχύσεων προς άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δε ότι κάποιοι από τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο ζουν σε χώρες μέσου εισοδήματος αυτή τη στιγμή. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση όποιων περιορισμένων πόρων ε, έχουμε στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειες και όχι μόνο να κάνουμε την ε, προσθετικότητα. Τώρα, γιατί έχουμε αναπτύξει επίσης κοινές προδιαγραφές για κοινέ δημοσιεύσεις και αυτό ήδη συμφωνήθηκε στον Μπουσάν όταν δημιουργήθηκε η διεθνής εταιρική σχέση. Τώρα, κατά πόσο το ΝΤΑΚ είναι το καλύτερο χώρος, το καλύτερο βήμα, ε, δεν νομίζω πως έχουμε και εναλλακτική όσον αφορά τη μέτρηση του, της επίσημης αναπτυξικής βοήθειας. Τα σώματα του, ε, του ΟΗΕ είναι πιο θεμητά, αλλά υπάρχει ένα παζάρεμα ανάμεσα στην θεμητότητα, την νομιμότητα και την εμπειρογνωμοσύνη. Και νομίζω πως έτσι αυτά τα θέματα μπορούν καλύτερα να συζητηθούν στο ΤΑΚ. Τελικό σχόλιο, υπάρχει μια σύσταση για την ατζέντα, για την αλλαγή και την συνένεση της Ένωσης για την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε πραγματικά να συμφωνήσουμε νομίζω με τη μελέτη εκεί όπου λέει ότι τόσο η συνένεση όσο και η ατζέντα για την αλλαγή δεν λαμβάνουν πραγματικά υπόψη την εξέλιξη στις συζητήσεις για την ανάπτυξη. Νομίζω πως σαφώς λέει τόσο στο κονσένσους όσο και στην ατζέντα για την αλλαγή αλλά και στην ανακοίνωσή μας όπου, που τιτλοφορείται ε, αξιοπρεπή ζωή για όλους μετά το 2015, ότι θέλουμε καθολική και βιώσιμη ανάπτυξη και όχι οποιοδήποτε είδος ανάπτυξη. Αυτές είναι οι βασικές μας παρατηρήσεις. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. το, του σβήνει το μικροφωνό της η Πρόεδρος. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γουάκενμπος που έχει πολύ δύσκολο επίθετο από την Concord. Πέντε λεπτά έχετε παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά, καλωσορίζουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την έκθεση, τη μελέτη αυτή και θεωρούμε και εμεί ότι είναι πολύ επικαιρή. Και θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε όσο πιο πολλέ απόψει γίνεται για την βέλτιστη δυνατή προσέγγιση στο μέλλον. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι στην ε, μελέτη όπου γίνεται λόγος για το, έργο της Concord Aid Watch. Καλύπτεται και από άλλες task forces. Εμείς καλύβουμε αυτά που εντάσσονται στα πλαίσια της επίσημας αναπτυξιακής βοήθειας, όχι αυτά που θα πρέπει να συμπληρωθούν. Αλλά προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μία συνένεση σε ό,τι αφορά την βέλτιστη δυνατή μεταρρύθμιση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές ροές και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, εδώ θα διαφωνήσουμε γιατί ανησυχούμε και είμαστε κάπως διστακτικοί. Είναι ύποπτη η προστατικότητα και πολλές από τις μεθόδους θα πρέπει να τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά προτού τις διαμορφώσουμε με σωστό τρόπο και επίσης δεν είναι πάντα πραγματικές ροές από ιδιώτες, από δωρητές στις χώρες που χρήζουν βοήθειας όπως για παράδειγμα στις εγγύησεις να υπογραμμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία. Συμφωνούμε με πολλά από τα πορίσματα της μελέτης, αλλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε τους τομείς εκείνους όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση χωριών πόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις, ε, για τις χώρες αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο φορολογικά ζητήματα, αλλά και κινητοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εταιριών σε εθνικό επίπεδο και στις ε, χώρες εταίρους. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε περαιτέρω για να είναι και πιο διεντελογικά και πιο αποτελεσματικά τα φορολογικά συστήματα και τις αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά τις ε, λοδαπές ροές. Δεν είμαστε κατά των ροών αυτών, αλλά να μην αντικαθιστούν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια αυτές οι ροές. Ακούσαμε διάφορα για τη νέα πραγματικότητα, αλλά είναι γεγονός για 37 χώρες η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι 10% των δαπανών του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό αυτό σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της κοινοφελής, την παιδεία, την επίδεξη των ε, δεσμεύσεων. Και Πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτές τις ευρύτερες ροές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, να περάσουν από εξέταση, να είναι διαφανείς, εύκολα στη μέτρηση και να έχουν σαφή συμπληρωματικότητα. Θέλει η Επιτροπή συνέργειες βασικά μας είπε, αλλά εμείς θέλουμε συμπληρωματικότητα γιατί υπάρχουν πολλές αλληλεπικαλύψεις. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ε, ε, συμβατικών χρηματοδοτήσεων, όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Και εδώ πέρα λοιπόν ε, αναπτύσσουμε στο φυλάδιό μας ε, τις αρχές αυτές. Συμφωνούμε με πολλά από τα ευρήματα της μελέτης και της έρευνας. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αναπτυξιακή βοήθεια <clears throat> χωρίς κάποιο αποτελέσμα σκοπό και αποτελέσμα στόχο. Και Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προτιμούμε αυτές τις μεθόδους, να μην βασιζόμαστε σε χρέο. Σε ό,τι αφορά την ε, μεγέντηση της ε, βοηθείας, θεωρούμε λοιπόν τα έξοδα για τους φοιτητέ, τα διοικητικά έξοδα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε πολύ σαφείς ε, προτάσεις για το τι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί μετά την ε, ε, μεταρρύθμιση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Και τέλος, να πούμε ότι ο ECD έχει μεν, έχει μεν τις δυνατότητες και τις ικανότητες, αλλά δεν έχει την νομιμότητα. Συνήθως τα πράγματα είναι ανάποδα είναι αντίστροφα. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να ε, καλύψουμε ένα ευρύτερο ε, φάσμα χρηματοπιστωτικών ορών και νομίζω ότι έτσι καλύπτουμε ε, τους πιο πολλούς τομείς τους οποίους θα θέλαμε να τονίσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαιρόμαστε που γίνεται αυτή η συζήτηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα επειδή η πόροι που θα προκύψουν από τη συζήτηση αυτή Ενδεχομένω να είναι αυτοί που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε του ε, αναπτυξιακού μα στόχου. Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στο μέλλον οι φυστάμενε δεσμεύσει. και να ε, σημειώσουμε ότι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε νέοι πόροι θα πρέπει να αποτυπώνουν και να σέβονται τους, ε, τις ήδη ανελημμένες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουάκενμπος. Έτσι είναι το όνομά σας, έτσι προφέρετε. Ναι, Κουάκενμπος, ναι. Είδα τι σου είναι ένα όνομα. Τώρα, θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Ο κύριος Κορτές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, το θέμα αυτό είναι κέριο και πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Μάλιστα έπρεπε να το είχαμε ήδη ε, συζητήσει, γιατί σχεδόν έχει διεκπαιρεωθεί η συζήτηση και κρίμα που δεν ε, εγκύψαμε στο θέμα αυτό πιο νωρίς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα με αυτά που είπα προλαλή σα. Και το έχουμε πει και διατρανώσει σε διάφορες συζητήσεις. Νομίζω ότι διανύουμε μια ιστορική στιγμή σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και την βοήθεια για τη συνεργασία. Και θα πρέπει να ετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορική αλλαγή, κυρίως με την ε, έλευση κάποιων καινοτόμων ε, ε, μορφών χρηματοδότησης. Γιατί η ιδιωτική χρηματοδότηση θα συνοδεύσει την δημόσια χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα συνεργασίας. Είναι πραγματικά ρηξικέλευτη αυτή και ιστορική στιγμή στην αλλαγή της αναπτυξιακής βοήθειας και της βοήθειας συνεργασίας. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Κονκόρτ. Θα πρέπει αυτά τα ιδιωτικά κονδύλια που ε, εντάσσονται στην αναπτυξιακή βοήθεια να διέπονται από τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συγκεκριμένη αξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί μπορούμε ε, αυτά τα καινοτόμα μέσα να τα συμπεριλάβουμε σαν να μην συνέβαινε τίποτα, αν και είναι όντως ε, περίεργο αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά, δεν έχω από τίποτα κατά ε, τη συμπερίληψη και ιδιωτικών κεφαλαίων στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει τα ιδιωτικά αυτά κονδύλια να υπάγονται σε συγκεκριμένους κανόνες και κυρίως να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Γιατί η συμπερίληψη των νέων ιδιωτικών κονδυλίων στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να διέπεται από τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και από σαφή αξιολόγηση και έλεγχο γιατί αυτό ζητούν οι πολίτες. Αλλιώς ε, θα έχουμε μία αλλαγή από την κερκόπορτα της επίσημης αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Χρειαζόμαστε αυτά τα ιδιωτικά κονδύλια σίγουρα για να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά επαναλαμβάνω και θα το κάνω συνεχώς, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη απόλυτη διαφάνεια και συγκεκριμένη σαφή αξιολόγηση για αυτά τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα συμπεριληφθούν στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ούτως ή άλλως τέτοια διαφάνεια και έλεγχο ζητούσαμε και για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, για τα δημόσια δηλαδή, τα κρατικά κονδύλια. Η διαφάνεια είναι το κέριο και πιο σημαντικό ζήτημα. Αυτά. Δεν μου άρεσε και πολύ ε, κάτι που είπατε για το τρίτο σημείο. Μεταξύ των προτεραιοτήτων ε, του συνεκτικού συστήματος ε, χρηματοδότηση αναφέρεται κάτι που δεν το πολύ κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό το έχει κάνει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που περιμένω από την έκθεση δεν είναι μόνο να μας πει τι θα πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενταχθεί στην όλη διαδικασία, αλλά τι θα πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιβληθεί η διαφάνεια ώστε αυτή η νέα μορφή που θα λάβει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη διαφάνεια. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή τη μέγιστη διαφάνεια για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Ώστε αυτό το νέο άλμα που θα γίνει, που θα είναι ιστορικού χαρακτήρα, γιατί πήγαμε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο στη συνεδρίαση για την, για την εξέλιξη των αναπτυξιακών στόχων και όλοι μας είπαν ότι το κέριο σημείο αυτή τη στιγμή στην ε, παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια είναι η συμπερίληψη ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης ε, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και μερικές φορές δεν γίνεται σωστή διαφοροποίηση μεταξύ του ιδιωτικού, των ιδιωτικών κονδυλίων και των δημόσιων. Εγώ είμαι υπέρ μιας συντονισμένης ε, και διαφανούς προσέγγισης με πρωταρχικό στόχο αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι η βασική μας μέλημα και μέλημα. Να βοηθήσουμε τις χώρες αποδέκτες που χρειάζονται αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί δεν θα πρέπει η εισαγωγή των ιδιωτικών κονδυλίων στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να είναι ένας λανθάνων τρόπο ή ένας έμεσος τρόπος για να επηρεάσουμε κοινωνικά μοντέλα ανάπτυξης στις χώρες αυτές. Η βοήθεια θα πρέπει να έχει στόχο τη βοήθεια των χιλιάδων ανθρώπων που τη χρειάζονται. Γι' αυτό θα πρέπει διαφάνεια να είναι το κύριο μας μέλημα. Γιατί είναι ιστορική στιγμή και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξίζει καλύτερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε πώς ακριβώς ε, θα συμπεριληφθεί αυτή η ιδιωτική χρηματοδότηση και η εισαγωγή των ιδιωτικών κονδυλίων στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και να έχουμε και τα πρώτα στοιχεία για την αξιολόγηση αυτής της αλλαγής και αυτής της εισαγωγής. Δεν είμαι κατά καταρχήν της ιδιωτικής χρηματοδότησης, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει διαφάνεια, γιατί γινόμαστε μάρτυρες μια ιστορικής αλλαγής της έννοιας της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, δύο λόγια για την μέθοδο. Έχετε δίκιο που υπογραμμίζετε στη μελέτη σας ότι χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και εκτιμούμε την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Και διευκρινίζω ότι πρόκειται για δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή είναι μια έννοια αρκετά σαφής, που ορίζεται από τον ΟΣΑ και όσον αφορά τις πολιτικές προτάσεις που διετυπώσατε, δηλαδή την ακύρωση του χρέους, που δεν μπορεί να ενταχθεί στην εκτίμηση της δημόσιας ε, αναπτυξιακής βοήθειας, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, εδώ δεν μας λέτε τίποτα νέο, το έχουμε ήδη εισάγει αυτό στην ε, μελέτη, ε, για, στο ενέκθεση μάλλον, για την μελλοντική αναπτυξιακή βοήθεια, έγινε δεκτό γενικά από το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, πρόκειται για διόρθωση των δικών μας λαθών. Πρέπει να είναι επιπλέον χρήματα. Δεν έχει σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Είχαμε μια πολύ αρκετά δυσάρεστη συζήτηση εδώ με την αρμόδια επίτροπο για το περιβάλλον και για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και επιμείναμε στη θέση μας. Για τη μέθοδο λοιπόν συμφωνώ. Η πολιτική μου παρατήρηση εδώ είναι ε, να δούμε πώς πρέπει να εκτιμήσουμε τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν ε, την, το επίπεδο το αναπτυξιακό των χωρών. Θέλουμε να προωθήσουμε διάφορο, τον ιδιωτικό τομέα, θέλουμε να προωθήσουμε τους μη κρατικούς φορείς, πολύ ωραία, άρα πρέπει ένα άλλο μέσο να υπάρξει και άλλα μέτρα για να εκτιμήσουμε τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Εδώ φυσικά ε, πρόκειται ε, για μια άλλη ένα άλλο σύνολο μέσων που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και όσον αφορά το Ινστιτούτο Διαφάνειας, νομίζω ότι πολύ εύκολα υποκύπτουμε στον πειρασμό της δημιουργίας νέων Ινστιτούτων όλη την ώρα. Εμείς εδώ αγωνιστήκαμε για να φτιάξουμε ένα Ινστιτούτο για την αναπτυξιακή βοήθεια, το οποίο θα μπορούσε διοικητικά να είναι συνδεμένο με την Κομισιόν, γραμμένοντας αμερόληπτο στην προσέγγιση του, δεν καταφέρουμε να το επιβάλλουμε, αλλά αυτό λείπει. τώρα ένα Ινστιτούτο διαφάνεια θα ήταν ένα παρατηρητήριο βασικά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτιμούμε την εξέλιξη των νότιων χωρών. Ε, οι ίδιες θα πρέπει να κάνουν μια πρώτη αξιολόγηση, να εκτιμήσουν σε ποιο βαθμό είναι το σύστημά τους διαφανές, ε, εάν η κοινωνία ή των πολιτών τους είναι αρκετά καλά δομημένη ώστε να αποτελέσει το αντίβαρο στην πολιτική να εκτιμήσουν αν τα κοινοβούλια τους είναι σε θέση να χειριστούν την δημοσιονομική διαδικασία. Οπότε νομίζω πως δεν τονίζεται αρκετά ο χειρισμός του του μέλλοντος από τις ίδιες τις ε, χώρες παραλήπτες, αποδέκτες της βοήθειας. Ε, το είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για κάθε είδους αναπτυξιακή βοήθεια και έπειτα ε, είπα, δημόσια βοήθεια, κλίμα, πρόσφυγες, όπου στον κατάλογο της βοήθειας, αναπτυξικής βοήθειας, είναι μια επίκριση που απευθύνεται στα κρατημέλη. Τα κρατημέλη είναι όσα. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν καλύπτεται από αυτές τις κριτικέ. Το θέμα για την Κομισιόν και για το Ευρωκοινοβούλιο και για την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι να καταφέρουν τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν στην άποψή του. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δανείζει τίποτα, τουλάχιστον όχι η Κομισιόν, άρα δεν έχει να, ανακτη... να κυρώσει κανένα χρέο. Μια τελευταία παρατήρηση είναι οι υποτροφίες και ο πολιτισμός. Πολιτισμός δεν είναι μόνο το φαΐ, η μάσα, να γεμίζουν τα στομάχια, είναι και να αναπτύξουμε προσωπικότητες. Και άρα λοιπόν ο πολιτισμός είναι κομμάτι του ανθρώπινου, της ανθρώπινης ανάπτυξης δεν υπάρχει θέμα λοιπόν να διαγραφεί αυτό από την αξιολόγηση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας στην ανάπτυξη. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις υποτροφίες ή την ε, χρηματοδότηση των υποτροφιών που έχουν αναλάβει τα κράτη δωρητές. Είναι μια επιχείρηση προώθηση ενός πολιτισμού ή μια συμμετοχή σημαντική στην ανάπτυξη μιας χώρας. Εάν χρηματοδοτήσετε μελέτες ε, ένα Σενεγαλέζου για παράδειγμα να γίνει γιατρός και μετά αν πάει πίσω να βοηθήσει τη χώρα του με τις γνώσεις του, μα αυτό είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί προς το συμφέρον της ανάπτυξης μιας χώρας εταίρου. Αν χρηματοδοτήσουμε τον φίλο του και αυτός εγκατασταθεί εδώ στην Ευρώπη, ε, τότε δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι απλά τα πράγματα. Χωρίς να δίνουμε υπερβολικά μεγάλη σημασία στα μέσα και στη μέτρηση αυτών, να κάνουμε σε κάθαρη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που βοηθά προφανέστατα στην ανάπτυξη και εκείνο που φαίνεται να βοηθά, ενώ στην πραγματικότητα δεν βοηθά. Ε, ε, Δίνω τώρα το λόγο στον, κύριο Πέντρο Μονασάνα. Sí, eh, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Μόνο δύο λεπτά δυστυχώς έχετε στη διάθεσή σας. Πάει και το ένα ήδη, ε, το ένα λεπτό εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι αυτό που κατέδειξε η σύντομη συζήτηση είναι η κατάσταση των πραγμάτων, η κατάσταση μάλλον των συζητήσεων. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Κορτές και συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά τα θέματα που έπρεπε δεν είχαν συζητηθεί. Πάντως η μελέτη αυτή κυρίως ευστά την προσοχή σας σε τρεις πιθανές ψεύδο εναλλακτικές λύσεις που είναι σημαντικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί το να πρέπει κανείς να διαλέξει μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης αναπτυξιακής βοήθειας είναι ε, ψευτοδήλημα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και οι δύο πλευρές είναι χρήσιμες. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε ούτε την ε, κρατική, τη δημόσια, ούτε την ιδιωτική χρηματοδότηση. Ούτε είναι απαραίτητο να διαλέξουμε μεταξύ της δωρεάς και του δανείου, γιατί πολλές φορές ε, η συμβολή ενός δανείου είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία ή την ε, χρησιμότητα μιας δωρεάς, ιδιαίτερα όταν αυτή φτάσει στα χέρια διεφθαρμένων πολιτικών και δεν φτάσει στους αποδέκτες. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ε, κύριε Γκέρενς, το πρόβλημα δεν είναι αν μια υποτροφία ε, για σπουδές ε, κάποιο που δεν είναι από τα πιο φτωχά στρώματα των χωρών είναι καλό ή κακό για την ανάπτυξη. Γενικώ μια υποτροφία είναι θετική και πολλές φορές είναι καλύτερη η χρηματοδότηση μιας υποτροφίας ε, γιατί ε, μπορεί να μένουν στην πλούσια χώρα οι φοιτητέ, όπως η δική μου περίπτωση. Το θέμα είναι ότι μερικέ χώρε χαρακτηρίζουν αυτή το τη δαπάνη ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και άλλες δεν το κάνουν. Μερικές ε, δηλώνουν ε, τις ε, δαπάνες αυτές ως τις βοήθειες στους πρόσφυγες ως αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ άλλες χώρες το κρίνουν αυτό ανήθικο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η απόφαση να δηλώσει κανείς την αναπτυξιακή βοήθεια είναι να πόκεται σε διακριτική ευχαίρεια του δωρητή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάος την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία για να μην διακυβευτεί η αξιοπιστία και η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη έχει κυλιδωθεί στον τομέα αυτό. Η συζήτηση είναι ανοιχτή. Ακούσαμε τις κριτικές ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα, τους ευνοϊκούς όρους των δανείων και γίνεται συζήτηση για αυτούς τους ευνοϊκούς όρους των δανείων κύριε Πράντα και η θέση του ΟΣΑ όπως φαίνεται στο άρθρο του Μάνινγκ στους Financial, Financial Times, ε, φαίνεται από εκεί ότι και τα ευνοϊκά δάνεια ε, υπάγονται σε πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς και ο καθένας τερμινεύει με το δικό του τρόπο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε διλήμματα όμως και να δούμε ποια είναι η κατάλληλη δομή που αντικατοπτρίζει καλύτερα και συμπεριλαμβάνει όλα τα μεμονωμένα στοιχεία και τις μεμονωμένες πτυχές της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Και νομίζω ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι αυτός που αναφέρεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας στην Ευρώπη είναι η εξάλληψη της φτώχειας και η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των φτωχότερων χωρών. Αυτό κατοχυρώνεται από την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας και με αυτόν τον προσανατολισμό και με αυτό, το, αυτή, με αυτό το, την αρχή ως πηξίδα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε μεγαλύτερη τάξη στην κατάσταση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Γουστάβο Μαρτίν Πράντα. Ε, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή καταδεικνύει ότι Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και περίπλοκα. Και γι' αυτό καλωσορίζουμε τη συνέχιση της συζήτησης και στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουμε επί ενός καινούργιου πλαισίου και ενός καινούργιου χρηματοδοτικού πλαισίου. Δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια να κάνω για τις παρεμβάσεις που ακούσαμε, να αναφέρω ότι συμφωνούμε με τη σημασία της διαφάνειας που τονίστηκε. Κάθε φορά που υπάρχει παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τη βοήθεια αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε νομίζω τη σημασία της διαφάνειας. Τώρα, η συζήτηση αυτή και τα σχόλια του κυρίου Γκέρενς οι χώρες δικαιούχοι θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα παρακολουθούν την χρήση των πόρων και των κονδυλίων που φτάνουν στις χώρες τους. Και αυτό νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνος όλους. Αποτελεί μία από τις μεγάλες αλλαγές που εισαγάγαμε στον Μπουρσάν όταν και ε, δημιουργήσαμε αυτή την παγκόσμια εταιρική σχέση και όποτε και συμφωνήθηκε ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πόρων θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο χώρας. Και αυτό νομίζω ε, ότι συμφωνήθηκε και στο Μεξικό. Ελπίζουμε μάλλον στο Μεξικό να είναι πολύ ενδελεχής η ανάλυση για την χρήση και τη διοχέτευση των πόρων ανά χώρα. Νομίζω για το θέμα των, ε, των προνομιακών δανείων. Όντως αληθεύει ότι δεν είναι απόλυτα σαφείς οι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό ισχύει. Αλλά κατά το παρελθόν η γραμματεία του ΝΤΑΚ έχει εφαρμόσει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές με διαφορετικό τρόπο για τους διαφορετικούς και γι' αυτό λοιπόν τα έχουμε θέσει υπό αμφιβολία, υπό αμφισβήτηση τα στοιχεία αυτά, τις κατευθυντήρες αυτές τις γραμμές. Συμφωνώ λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τον ορισμό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε από έναν οργανισμό που ελέγχει τις χρηματοπιστωτικές ροές είναι να εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια για τους δωρητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και δίνουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κουάκενμπος. Uh, Σας ευχαριστώ. Δεν έχω και εγώ πάρα πολλά να προσθέσω. Συμφωνώ απόλυτα ότι η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πιστεύω επίσης ότι από εκεί πηγάζει και η αξιοπιστία και η κριτική αξιολόγηση ιδιαιτέρως των, ε, ε, των ιδιωτικών ροών που μπορεί να στρεβλώσει το εσωτερικό των χωρών. Για τα υπόλοιπα σχόλια δεν έχω ιδιαίτερα να προσθέσω, ιδιαίτερα πολλά να προσθέσω, αλλά πολλά από τα μέσα που χρησιμοποιούνται πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάνουν το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι προσπαθούν να πετύχουν και ποια είναι η χρησιμότητα του να δημιουργηθεί ένα καινούριο μέσο τη στιγμή που υπάρχει ένα ήδη εφιστάμενο μέσο που λειτουργεί αποτελεσματικά ενδεχομένως. Άρα, θα πρέπει κυρίως να κοιτάξουμε την αποτελεσματικότητα και όχι το κατά πόσον κάτι είναι καινούριο, αλλά φυσικά να εξετάσουμε και τα νέα αυτά μέσα, εφόσον η μεθοδολογία για την αξιολόγησή τους είναι αξιόπιστη. Τέλος, η συζήτηση για τα προνομιακά δάνεια είναι ένας από τους τομείς που προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού γιατί εμπλέκονται, ξέρετε, και τα επιτόκια. Τα κίνητρα δε για τις ε, οργανώσεις παροχής βοήθειας είναι μεγαλύτερα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο δεν ανταμείβει τις χώρες που εστιάζονται στην βοήθεια την αναπτυξιακή. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή μια δομή κινήτρων που θα εστιαστεί σε αυτά τα σε αυτές τις ε, πτυχές, ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλες ανάγκες για υπηρεσίες κοινοφελής. Είναι λοιπόν σημαντική η συζήτηση αυτή και για διάφορους λόγους επί μακρόν η όλη η συζήτηση δεν είχε εστιάσει την προσοχή του κοινού. Ελπίζουμε μέχρι το Δεκέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή ή έστω μέχρι το Μάρτιο. Είναι λοιπόν πολύ επικαιρία αυτή η μελέτη αυτή η έρευνα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τι συζητιέται, Ποιε θα, είναι οι επιπτώσει για του πόρου, γιατί αυτό θα έχει μεγάλε συνέπειε για τη συζήτηση μετά το 2015. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Α περάσουμε τώρα σε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων για τι τροπολογίε που υποβλήθηκαν για τη γνωμοδότηση του κυρίου ε, Γκερέρου και που αφορά την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της στην συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή που είναι αρμόδια από τις ουσίες είναι η ΑΦΕΤ ε, και η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται σε μια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δυστυχώς ο κύριος δεν είναι εδώ, ο κύριος Γκερέρο. Δεν μπόρεσε να έρθει στη σημερινή μας συνεδρίωση. Allora, ah, ecco bene. Prende la parola. Θα λάβει στη θέση του το λόγο ο κύριος Χόρτες Λάστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ εδώ ο κύριος Γκερέρο. Μου ζήτησε όμως να σας παρουσιάσω εγώ τα συμπεράσματά του. Θα σας διαβάσω λοιπόν το έγγραφο που μου έδωσε. Στις 11 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πατεκπρόσωπος ε, έδωσαν την κοινή ανακοίνωση για την ε, προσέγγιση της, ε, γενική προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για το χαρακτηρισμό μιας στρατηγικής που συνδυάζει την ανάπτυξη με άλλα, όργα, με εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής. Και αυτή η ανακοίνωση για την συνολική προσέγγιση της εξωτερικής δράσης αποτελεί την ευκαιρία για να διευκρινίσουμε και να κάνουμε πιο λειτουργική την ε, προσέγγιση σε, στην περίοδο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, στόχος της ανακοίνωσης είναι να χρησιμοποιήσει όλες τις πολιτικές και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν ε, τη διπλωματία, την ασφάλεια, την άμυνα, το εμπόριο, τα χρηματοπιστωτικά θέματα, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν κάποιες κρίσεις στο εξωτερικό. Οι ιδιαίτερα σημαντικέ είναι του κυρίου Πρέντα, το ΕΛΚΑ και μπορεί ο εισηγητής να να συμφωνήσει. Είναι σημαντικό σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια της συνολικής αυτής προσέγγισης. Θα πρέπει επίσης να καλύπτονται όλες οι φάσεις ε, της σύγκρουσης, από την έγκαιρη προειδοποίηση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση της κρίσης, ε, διαχείριση της κρίσης, αποκατάσταση τη κατάσταση και της ειρήνης. Δεύτερον, αναφέρονται οι ιδιαίτερες αρχές της αναπτυξιακής ε, και ανθρωπιστικής βοήθειας και επίσης ε, ε, αναλαμβάνει τη δέσμευση, μακροπρόθεσμη δέσμευση υπέρ της ειρήνης, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας ό,τι αφορά την τον κίνδυνο να μην επικρατήσουν μόνο οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής επί των στόχων της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Εμείς ε, ως Επιτροπή ανάπτυξη, θα πρέπει να τονίσουμε την πιθανή ένταση που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ τη ε, συνοχή των ε, αναπτυξιακών πολιτικών αφενό και τη συνολική προσέγγιση διαχείριση των κρίσεων εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. βασικό στόχο τη αναπτυξιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξάλληψη τη φτώχεια, ε, οπότε είναι σημαντικό ο στόχος κατα... της τη της να μείνει στο περιθώριο της, να πολιτική εξωτερικής και η συνολική αυτή προσέγγιση να μην διαβρώσει τον πολιτικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής πολιτικής βοήθειας. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα προγράμματα ασφάλειας να μην παρεμποδίσουν το προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η ανθρωπιστική βοήθεια να υπηρετεί πολιτικού σκοπούς ή να θεωρείται εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων. Επίση, για να είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση σε πληθυσμού που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, η βοήθεια αυτή δεν πρέπει μόνο να είναι ουδέτερη, αλλά και να φαίνεται ω τέτοια. σε λίγο θα γίνει και η ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης αυτής και ο συντάκτης ευχαριστεί τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Ο κύριος Πόγκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου είναι μια ε, παρέμβαση του κυρίου Πρέντα που είναι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ και που αυτή τη στιγμή επιστρέφει από το Κόνακρι, όπου παρουσίασε τη τελική έκθεση των παρατηρητών των εκλο... της εκλογικής διαδικασίας εκεί. Ε, είναι πρόεδρος μάλιστα της Αρμόδιας Επιτροπής ε, για την Επίβλεψη των Εκλογών. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ για την έκθεση αυτή μας επέτρεψε να εξετάσουμε καλύτερα τις εξωτερικές επιπτώσεις της συνολικής προσέγγιση Ένωσης. Είναι αλήθεια πως η συνολική προσέγγιση είναι νέα έννοια που τώρα παγιώνεται στην Ένωση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε εξ αρχή τη τακτική. Αντίθετα, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία ώστε να εξασφαλίσουμε πω οι θέσει μα θα ληφθούν υπόψη στη διατύπωση τη σφαιρική συνολική προσέγγιση. Ο κ. Πέντα συμφωνεί απόλυτα πω η συνοχή στο πλαίσιο τη συνολική προσέγγιση δεν θα πρέπει να σημάνεται κυριαρχία των στόχων των εξωτερικών πολιτικών επί των αρχών τη αναπτυξιακή συνεργασία και της ανθρωπιστικής δράσης την οποία υπερασπίζει η Επιτροπή μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουμε ότι η κοινή ανακοίνωση για τη συνολική προσέγγιση την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το Δεκέμβριο του 2013 περιλαμβάνει αρκετές πρόοδους. Ας πούμε γίνονται σαφείς αναφορές στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι αρχές της αναπτυξιακής βοήθειας και της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης τονίζονται η πρόληψη των συγκρούσεων και η λήψη υπόψη ε, του, του απότερου μέλλοντος. Ε, για τον κύριο Πρέντα, βασική θέση της συνολικής προσέγγισης, βασικό θέμα μάλλον θα είναι η πρακτική εφαρμογή της συνολικής προσέγγισης και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτή θα βασίζεται σε κοινέ αναλύσεις και σε κοινέ πληροφορίες τις οποίες θα μοιράζονται τα διάφορα όργανα που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία και επίσης από μια σαφή κατανομή των ευθυνών. Αν θέλουμε πραγματικά να είναι λειτουργική η συνολική προσέγγιση, θα χρειαστούν κατευθυντήριε γραμμές για την εφαρμογή της και η εφαρμογή της θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τακτικών εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Ταυτόχρονα χρειάζεται ε, σαφής δέσμευση από την ΥΠΑΤΕ εκπρόσωπο και από την Κομισιόν θα εξασφαλίσουν τη συνοχή των εξωτερικών σχέσεων σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης ε, της εξωτερικής επιρροής των πολιτικών μας. Αυτά είναι και τα θέματα των εννέα τροπολογιών που έχει υποβάλει ο κ. Πρέντα εξ ονόματος του ΕΛΚΑ και ελπίζει πως οι και οι σκιώδες εισηγητές των ομάδων θα μπορέσουν να τη στηρίξουν. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κ. Πόγκα και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης αλλά και τον κύριο Κορτές Λάστρα που αναπλήρωσε εδώ τον εισηγητή. Το σημείο που με ενδιαφέρει κυρίως ε, στη γνωμοδότηση δεν είναι κάτι το απτό, γιατί η σύγκρουση που αποφεύθηκε δεν φαίνεται πουθενά. Οπότε πώς θα εξάρουμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κανένας δεν έλαβε Νόμπελ Ειρήνης για πόλεμο που αποφεύχθηκε, που κατάφερε να τον προλάβει και τελικά δεν εκτελήχθηκε. Μία επιτυχής ε, εκλογική διαδικασία που επιτρέπει την ε, καλύτερη διακυβέρνηση, τη μετάβαση στη δημοκρατία. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα της ε, εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει σε μια τέτοια κατάσταση. Εγώ είμαι υπέρ της εξωτερικής δράσης ε, και θα ήθελα να είναι πιο παρούσα η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φαίνεται σε τομεί όπου δεν εξασφαλίζεται κατά απαραίτητα η ορατότητα, αλλά που υπάρχει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στο διεθνές προσκήνιο. Οπότε Έχουμε μεγάλη πρόοδο στην επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δυστυχώς μεγάλη αδυναμία στην προβολή αυτής της πολιτικής και των πλονεκτημάτων της. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα. Ε, πώς θα αποφύγουμε, θα παρεμποδίσουμε μια γενοκτονία. Η, το πλωστάσιο μας ε, των εργαλείων και των μηχανισμών της της εξωτερικής πολιτικής και της ε, διεθνούς πολιτικής ε, μπορεί να αποτρέψει γενοκτονίες σαν αυτή που έγιναν στη Ρουάντα για παράδειγμα. Για να έχουμε διάφορα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, συναγερμού. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά εργαλεία στον κόσμο για να ενημερωνόμαστε έγκαιρα για κάποιες έκρηθμες καταστάσεις και να αποτρέψουμε τραγωδίες. Θα μπορούσαμε να επιμείνουμε λοιπόν στην πολιτική δράση. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα του βαθμού συμμετοχής των κρατών μελών. Γιατί αν η Γαλλία δεν είχε δώσει το παρόν στο Μάλι, θα ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση στη χώρα αυτή. Το ίδιο ισχύει και για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. μία χώρα στέλνει στρατιώτες, άλλη νοσηλευτικό προσωπικό. Γίνεται ένας επιμερισμός ε, των ε, καθηκόντων, αλλά στο θέμα αυτό νομίζω χωλαίνει πολύ ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το δίκαιο καταμερισμό των ε, αποστολών και των καθηκόντων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ε.Ε. τον κύριο Σαν Λάρστρομ. Thank you very much, Madam Chair. And... Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ε, εργάζομαι στην ε, διεύθυνση της ε, Υπηρεσίας Εκτορικής Δράσης για την βοήθεια αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας καλέσατε εδώ για να μιλήσουμε για αυτή την συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί μία από τις, ένα από τα θέματα τα οποία συζητιούνται ιδιαίτερως και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον τύπο, στην κοινή γνώμη για το τι θα μπορούσε να πετύχει αυτή η συνολική προσέγγιση. Θεωρώ ότι αυτή η ιδέα της συνολικής προσέγγισης προέρχεται από την ίδια πηγή, όπως και άλλα θέματα. Το θέμα είναι να συνενωθούν λοιπόν εργαλεία και μέσα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας σε ό,τι αφορά και την ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε για μια ολική λοιπόν τέτοια προσέγγιση που θα συνενώσει τους πόρους και τα εργαλεία, τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά έχουν συζητηθεί και τέλος, όπως είπε η Πρόεδρος, είπα ότι εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο πέρσι παρουσίασαν μια σχετική ανακοίνωση και τώρα συνεχίζεται η συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Η κοινή ανακοίνωση και οι βασικοί στόχοι είναι γνωστοί σε όλους φαντάζομαι και είναι και εύκολοι στην κατανέωση τους. Καλύτερη συνεργασία, συνένωση ε, μέσων και πόρων για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα είναι αρκετά ε, πράγματα κοινή λογικής, να το θέσουμε έτσι βάσει κοινών αναλύσεων, όπως ανέφερε και ένας βουλευτής, με κοινέ στρατηγικές, κοινέ προσεγγίσεις, αλλά όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα, αλλά και από τα κράτη-μέλη και σε επιχειρησιακό και σε πολιτικό επίπεδο. Βασικά πρόκειται για μία μέθοδο, ένα τρόπο εργασίας, για μία προσέγγιση, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο τίτλος. Αλλά ασφαλώς δεν θα πρέπει εκεί να περιοριστούμε δεν είναι μόνο φιλοσοφική προσέγγιση, αφορά και τις συγκεκριμένες δράσεις. Τι μπορούμε να αλλάξουμε στον τρόπο δράσης μας. Και αυτό εν μέρει αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση. Ελπίζω και τα υπόλοιπα στοιχεία να ακολουθήσουν. Κάποια από τα πράγματα αυτά τα πραγματοποιούμε ήδη. Κάποια άλλα τα εφαρμόζουμε εδώ και καιρό, κάποια άλλα θα πρέπει να τα αναπτύξουμε περαιτέρω και όταν μιλώ σε πρώτο πληθυντικό εννοώ για τα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώ και οι υπόλοιποι φορείς. Το θέμα λοιπόν είναι να καταστούν λειτουργικά αυτά. Έχουν τεθεί κάποιε εξαιρετικέ προτάσει στη συζήτηση, τι οποίε και πολύ ευχαρίστω ε, θα ήθελα να ακούσω περαιτέρω. Αυτά επί του παρόντος και θα χαρώ ασφαλώς να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Κορτές, θέλετε κάτι να πείτε. Όχι. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω κάτι σημαντικό. Η ψηφοφορία θα γίνει το απόγευμα σήμερα. Τι ώρα είναι? 11. Ε, στις 3 θα γίνει η ψηφοφορία. Allora, eh, abbiamo ritrovato. Sì, <laughs> abbiamo perduto il foglio. Allora, cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μερίσια διάταξή μας τώρα προβλέπει μια σύντομη εκθεσή από την, ε, ε, την αποστολή παρακολούθησης των εκλογών του Ευρωκοινοβουλίου στη Μαδαγασκάρη. Θα ακούσουμε τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου. Η συνά... Ήταν η κυρία Μπουλόν, η Παρτήρηση των εκλογών λοιπόν εκεί ήταν, ήταν περίπλοκη γιατί πέρα από την αποστολή παρακολούθησης των εκλογών του Κοινοβουλίου βρισκόταν και μια αποστολή παρακολούθησης των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την οποία ε, οδηγούσε η συνάδελφος Μούνιθ Ρουκίσα. Και η αποστολή της ε, Ισομερούς Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, και Ε, της οποίας συμπροέδρευε ο συνάδελφος Τυρολιέν και ε, Φίτ Τζάκσον της Τζαμάικα, συμπρόεδρος της ε, Ισομερούς Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για το τμήμα κομμάτι ΑΚΕ. Ο κύριος Τυρολιέν μας ενημέρωσε ότι δυστυχώς επειδή βρίσκεται στη Γουαδελούπη δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συμμετέχει στην συνεδρία σήμερα και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπουλόμ στον κύριο Μπουλό με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εσείς είπατε ότι ε, η, η, η αποστολή, η παρακολούθηση των εκλογών, ε, εποπτείας των εκλογών ήταν ευαίσθητη. Όχι, δεν ήταν. Πολύ καλά πήγαν τα πράγματα. Η κυρία Άστον αποφάσισε να στείλει μια αντιπροσωπεία παρακολούθηση των εκλογών και η Προεδρία μας μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Ο συντονισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες ε, ανάμεσα στην κυρία Μουνής που ηγείται της ε, αποστολή παρακολούθησης και εμένα και των συναδέλφων ήταν εξαιρετική. Και τα σχόλιά μας ε, στις αντίστοιχες ε, συνεντεύξεις τύπου ήταν Παράλληλα, δεν υπήρχε πρόβλημα λοιπόν από αυτή την άποψη ούτε από την άποψη του συντονισμού. 120 παρατηρητέ είχαν έρθει από διάφορα κρατημέλη και αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη Μαδαγασκάρη Επίσης υπήρχαν παρατηρητές από την Ελβετία και από την Νορβηγία. Οι προεδρικές εκλογές λοιπόν αποφάσισαν στην πρώτη ε, γύρω για τις 25 Οκτωβρίου και ο δεύτερος για τις 20 Δεκεμβρίου και στις 20 προβλέπονταν και γενικές εκλογές ε, την ίδια μέρα. Ε, θυμίζω ότι στο πολιτικό πλαίσιο από το 2009 ο προηγούμενος πρόεδρος Μανάν εκδιώχθη από τον Ράζολιν και οι ε, διεθνείς οργανισμοί ε, άρχισαν διπλωματία για να προσπαθήσουν να φτάσουν στην εφαρμογή του φύλου πορείας που είχε συνυπογραφεί από όλους τους εκπροσώπους Μαδαγασκάρης, πολιτικά κόμματα κτλ. Και υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή του ε, γιατί αυτό σημαίνει και την διεξαγωγή αυτών των εκλογών. Μπορέσαμε με τη Διεθνή Επιτροπή να αποφύγουμε οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές της κρίσης, δηλαδή ο πρόεδρος ε, ο πρώην και ο μεταβατικός πρόεδρος να μην είναι υποψήφιοι, ωστόσο υπέβαλαν ο καθένας έναν υποψήφιο και μέσω εκείνων έγιναν εκλογές σχεδόν ε, ε, συγκαλυμμένες εκλογές έγιναν ανάμεσα σε δύο πρώην πρωταγωνιστές, οι οποίοι είχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία με 2 εκατομμύρια ευρώ για την δραστηριότητε τη ΕΛΕΤ και 15 εκατομμύρια για την εκλογική διαδικασία, χωρί να μιλήσουμε για το 1ο και 10ο φέντε που τα γνωρίζετε. Η αποστολή παρατήρησης ε, ήρθε σε επαφή με όλους τους φορείς, υποψηφίους της ΕΝΙΤ, ειδικό εκλογικό δικαστήριο και κοινωνία των πολιτών, ε, συναντήσαμε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο για να δούμε ποιες ήταν οι πιθανότητες απάτης στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας που θα διαρκούσε δύο μέρες. Όπως σας είπα, μιλήσαμε και για 120 παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν 5.000 ε, ε, και 10.000 αντίστοιχα παρατηρητές από την ίδια τη Μαδαγασκάρη στα 10.000 εκλογικά κέντρα. Ε, υπήρχαν παρατηρητές και από την Αφρικανική Ένωση και από την Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού, της και από τη Φραγκοφωνία. Ε, δεν παρατηρήσαμε να, υπάρξει καμιά, να υπήρχε καμιά στρέβλωση στις εκλογικέ διαδικασίες. Αυτό που κυρίως θέλαμε να καταγγείλουμε στα συμπεράσματά μας ήταν η απουσία δεν υπήρχε ανώτατο όριο για τις δαπάνες, τις εκλογικές δαπάνες, δεν υπήρχε διαφάνεια για τους πόρους. Οι δύο πρώτοι υποψήφοι λοιπόν που, που ε, αντιπροσώπευαν με τους δύο προηγούμενους πρόεδρους είχαν μια μέση παρουσία που ήταν γιγάντια. Όχι μόνο σε σχέση με το επίπεδο ζωής στην ζωή, στην Μαδαγασκάρη, γιατί οι κάτοικοι εκεί είναι συνηθισμένοι στο ότι δαπανώνται τεράστια ποσά για τις εκλογές, αλλά που ξεπεράστηκαν, ε, ε, ξεπεράστηκε κάθε όριο κυρίως από πλευράς του Προέδρου ΕΡ που ήταν ε, ο εκπρόσωπος του μεταβατικού Προέδρου και που νίκησε με μεγάλη διαφορά και που φαίνεται ότι χρησιμοποίησε πόρους κρατικούς εκτός που χρησιμοποίησε και ξένους πόρους που προέρχονταν δηλαδή από άλλες χώρες ίσως και από την Κίνα αλλά και που μπορεί να προέρχονταν από διαφθορά στην ίδια τη χώρα. Το θέμα λοιπόν της ουδετερότητας των μεταβατικών αρχών δεν αναφέρεται στον εκλογικό νόμο γιατί καθένας από τους πρώην προέδρους, ο πρώην πρόεδρος και ο μεταβατικός ε, αναμίχθηκαν στην εκστρατεία ενώ θεωρητικός δεν έπρεπε να συμμετέχουν στις εκλογικές συναντήσεις, στις προεκλογικές μάλλον συναντήσεις. το ειδικό εκλογικό δικαστήριο την παραμονή των εκλογών αποφάσισε να καταργήσει αυτή τη διάταξη ως διαμαγείας πριν από μια-δυο μέρες, ενώ είχε γίνει όλη η εκστρατεία ήδη. Οι δύο υποψήφοι λοιπόν ήρθαν ε, πρώτοι, οι δύο για τους οποίους μίλησα και μόλις ανακηρύχθηκε πρόεδρος ο ε, υποψήφιος του μεταβατικού πρόεδρου που ονομάζεται <laughs> Ερ, Ράτζα, Μουναπιανίν. Ε, τα ονόματα εκεί είναι συνήθως έτσι μεγάλα και ο αντίπαλος ζήτησε από την ΣΕΟΕΣ γίνει έρευνα για να τονιστούν οι ανομαλίες ε, που έγιναν στη διάρκεια της ε, εκλογική διαδικασίας. Πάντως, μέχρι στιγμής αυτό δεν μπορεί να αντιστρέψει το ποσοστό των ε, ψηφοφόρων και η ΣΕΕΣ εξετάζει τη δυνατότητα προσφυγής για αυτά τα εκλογικά κέντρα όπου υπάρχει διαμαρτυρία. Πάντως, τους ή άλλως δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. 61,5% υπήρχε συμμετοχή και 50% στο δεύτερο γύρο. Οι ε, γενικές εκλογές επίσης εξελίχθηκαν πολύ καλά. Ε, αυτό το κόμμα ε, του μεταβατικού πρόεδρου επίσης κέρδισε. Μένουμε δηλαδή στην ουσία στην ίδια πορεία, πράγμα το οποίο ελπίζω δεν θα είναι εις βάρος του πληθυσμού της χώρας. Αυτά συνοπτικά είχα να σας πω. Επαναλαμβάνω εκ νέου πως ο συντονισμός ανάμεσα στην ΑΚΕ ε, την ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, την ε, αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας. Οι ίδιες οι εκλογές έγιναν καλά και οι διορθώσεις τις οποίες είχαμε υποδείξει στον πρώτο γύρο ελήφθησαν υπόψη και για το δεύτερο γύρο και ότι οι μόνες ανομαλίες που καταγγείλαμε έντονα ήταν Αυτές που μας οδήγησαν να σκεφτούμε στο ότι υπήρχε χρηματοδότηση που προερχόταν από τη διαφθορά, δεν υπήρχε διαφάνεια στις δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία και ούτε και ανώτατο όριο. Αυτά. Ο, η επικεφαλής της αποστολής θα πρέπει να ε, επιστρέψει σε λίγο καιρό για να παρουσιάσει τα πορίσματά της και ε, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Θα είμαι λακωνικότατος. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μαρία Μονής για το εξαιρετικό έργο της ε, ως επικεφαλής της ε, Αποστολής Παρατήρησης των Εκλογών και να συγχαρώ και ολόκληρη την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί για μια ακόμη φορά έδειξε τον υψηλό επαγγελματισμό, το εξαιρετικό έργο σε μία ακόμη αποστολή παρατήρηση εκλογών. Πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν 120 οι πολιτικοί που μετέβησαν εκεί, το επιτελείο της παρατήρησης. Τώρα ανέκυψαν κάποιες υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Πάντως, στη τελική ανάλυση ήταν πολύ καλός ο συντονισμός με την Ισομερή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολύ σημαντικό να εμείνουμε στη θέση μας ότι σε τελικό βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίνει τη συνέντευξη τύπου και να δίνει την κοινή θέση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία της Μαδακασκάρης, γιατί ήταν τεράστιο το έργο σας και νομίζω ότι η επικεφαλής αντιπροσωπείας αυτής θα πρέπει να δίνει τη συνέντευξη τύπου. Γιατί έγινε μια απόπειρα και δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, είναι σημαντικό να μένει στεναρή στη θέση τη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνει μια συνοπτική ανακεφαλαίωση του έργου τη και να μην διατρέχουμε τον κίνδυνο τελευταία στιγμή να γίνει δήλωση που θα αποκλίνει από την γενική γραμμή του επιτελείου της παρατήρησης των εκλογών και αυτούς 120 ανθρώπους που τόσο σημαντικό έργο επιτέλεσαν καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής. Θερμά ευχαριστώ λοιπόν και στην κυρία Μουνίσα και σε την πολυμελή αυτή αντιπροσωπεία που για μια ακόμη φορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιζουά λέγομαι. Είμαι αρμόδιος για τη Μανταγασκάρη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπουλό, την ομάδα του και την κυρία Μουνίσα και τη δική της ομάδα για το εξαιρετικό του έργο καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής παρατήρησης ε, της εκλογικής διαδικασίας στη Μαδαγασκάρη. Γενικώ ε, συμφωνούμε με την πρώτη αξιολόγηση που έγινε και από την ε, αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που καταλήγει σε ένα σχετικά θετικό συμπέρασμα και αποτίμηση της διεξαγωγής των εκλογών. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της φιλοπορίας, το δικό της οδικό χάρτη για την εξομάλυση των ε, σχέσεων και τη συνεργασία μας με τη Μαδαγασκάρη και οι εκλογές αφενός, αλλά και κυρίως ε, η ανάληψη ε, του έργου των θεσμών που θα πρέπει να γίνει με αξιόπιστο τρόπο, αφετέρου θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες εξομάλυσης των σχέσεών μας με τη Μαδαγασκάρη. Περιμένουμε φυσικά την έκβαση ε, και την ε, δημοσίευση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, καθώς και την ε, συγκρότηση όλων των θεσμικών οργάνων, της, την Προεδρία, τη συγκρότηση σώμα της Βουλής, την, το σχηματισμό της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες εφόσον καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ήταν αξιόπιστες οι εκλογές. Και επέτρεψαν την ε, επαναφορά της χώρας ε, στη συνταγματική τάξη. Εφόσον λοιπόν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα θα ξεκινήσουμε μία σειρά ε, διαδικασιών προκειμένου με βάση το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού να επανέλθουμε στη εξομάλυση στο σχέσιο με την Μαδαγασκάρη. Βρισκόμαστε σε αναμονή, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση. Κύριε Μπουλόν, θέλετε να ευθερολογήσετε για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, και εγώ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο για τις ε, εξελίξεις ε, της πολιτικής κατάστασης στη Μαδαγασκάρη και την κατανομή του πλούτου της χώρας στον πληθυσμό. Και δεύτερον, θα ήθελα να σας μιλήσω για τον αντίκτυπο και την απήχηση που είχε η παρουσία της παγκόσμιας κοινότητας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τόπιο πληθυσμό κατά τη διεξαγωγή των εκλογών. Όπου και να πήγαμε, σε όποιο εκλογικό τμήμα και να πήγαμε και στο πιο μικρό, οι ντόπιοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους ε, προς την αποστολή μας για την ε, παρατήρηση των εκλογών. Και ευελπιστούμε ε, ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα συνεχίσουν και πάλι να ρέουν τα κοινοτικά κονδύλια και θα βελτιωθεί η κατάσταση του τοπικού πληθυσμού. Πάντως η παρουσία μας ήταν συμβολική και πολύ σημαντική για τον πληθυσμό της Μαδακασκάρης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση της UNICEF με θέμα την καταχώρηση των γεννήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως γνωρίζετε, η επίσημη καταγραφή ενός παιδιού τη στιγμή της γέννησης από πλευρά της κυβέρνησης αποτελεί το βασικό στοιχείο για την προστασία των πολιτικών, αστικών, οικονομικών και κοινωνικών του δικαιωμάτων. Μάλιστα, η εγγραφή του αποτελεί ένα είδος ε, διαβατηρίου για την προστασία από την εργασία των ανηλίκων, από τις πρόωρεους γάμους, από το εμπόριο και από τη ε, σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά αποτελεί και ένα στρατηγικό μέσο για κάθε κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να προγραμματίσει, να εφαρμόσει και να παρακολουθήσει τα μέτρα προστασίας. Το μεγαλύτερο τμήμα των μη εγγεγραμμένων παιδιών βρίσκεται στις πιο φτωχές χώρες, ιδιαίτερα στις περιοχές της ε, ε, Νότιας Αφρικής, ε, κάτω της Σαχάρας και στη Νότια Ασία, όπου τα μεσά παιδιά κάτω των 5 ετών δεν έχουν πιστοποιητικό γεννήσεως. Αυτή τη στιγμή περίπου 230 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών δεν έχουν ποτέ καταγραφεί. Και αυτό αποτελεί ένα πραγματικά ανησυχητικό σενάριο, ιδιαίτερα επειδή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ζουν σε χώρες όπου σοβούν ένοπλε σειράξεις ή εμφύλοι πόλεμοι. Και τώρα δίνω το λόγο στην Λίλα Πίτερς, εδώ, α, εσείς είστε, καλώς ορίσατε, της UNICEF για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή της για την εξέλιξη των γεννήσεων και να μας δώσει κάποιες υποδείξεις για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και λυπάμαι γιατί έχω κρυώσει, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μιλήσω καλύτερα. Η μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ σήμερα από πλευρά της UNICEF να παρουσιάσουμε την πρώτη ε, ολική συνολική ε, μελέτη για τις καταχωρήσεις γενέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά και πολύ γρήγορα θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα της ε, έκθεσης, της μελέτης. Βλέπετε λοιπόν στις διαφάνειες τι σημαίνει καταχώρηση γεννήσεων, το είπε η κυρία Πρόεδρος, δεν θέλω να απέκταθω, να υπογραμμίσω τρία πράγματα, ότι πρόκειται για τη διαρκή, μόνιμη και καθολική καταχώρηση των γεννήσεων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχιστεί και υποστηρίζουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να καταχωρίζουν τις γεννήσεις. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τις κυβερνήσεις και για τα ληξιαρχεία. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Σήμερα έχουμε 230 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών που ποτέ δεν έχουν καταχωριστεί σε ληξιαρχεία. Τα πιο πολλά εξ αυτών είναι στην Ασία. Ένα στα τρία δε ζει στην Ινδία. 57 εκατομμύριο, εκατομμύρια γεννήσεις σας ανέφερα, ή δεν σας τον ανέφερα μάλλον, ότι θα πρέπει να γίνεται από τις ε, αρχές της εθνικές η καταχώρηση. Τέσσερα από τα δέκα μωρά που γεννήθηκαν το 2012 δεν καταχωρήθηκαν. Δεν 57 εκατομμύρια. Σήμερα ένα στα 7 παιδιά που έχουν καταχωριστεί δεν έχουν ε, λεξιαρχική πράξη γεννήσεων. Γεννήσεως. Μπορεί να έχει καταχωριστεί δηλαδή το παιδί, αλλά να μην έχει λεξιαρχική πράξη γεννήσεως, γιατί συχνά οι γονείς δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα τέλη. γεννείται το παιδί δηλαδή, αλλά σε μεγάλη απόσταση από την σχετική ε, αρχή. Και έτσι η καταχώρηση αργεί και έτσι πολλά παιδιά σήμερα, 290 εκατομμύρια σήμερα παιδιά κατά των 5 δεν έχουν ε, ληξιαρχική πράξη γέννησης σε παγκόσμια κλίμακα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ε, πώς διαμορφώνεται στις διάφορες περιφέρειες η καταχώρηση των γεννήσεων και βλέπετε ότι βασικά ε, η Νότια Αφρική και η Νότια Ασία παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και στο ιστορικό της Αφρικής υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ένα χάρτη όπου αποτυπώνεται καλύτερα ε, που εστιάζονται τα προβλήματα. Έχουμε αριθμητικά στοιχεία για όλες τις χώρες. σας έχει δοθεί αυτή η μελέτη είναι πολύ σαφή τα στοιχεία. Αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να πετύχουμε μεγαλύτερη καταχώρηση των γεννήσεων, ξέρουμε που πρέπει να παρέμβουμε. Ένας άλλος, ένα άλλο θέμα είναι γιατί δεν καταχωρίζονται τα παιδιά που γεννιούνται. Κυρίως επειδή οι μητέρες συχνά δεν κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να καταχωριστεί η γέννηση του παιδιού τους και υπάρχει μεγάλη ε, σύνδεση μεταξύ της ε, παιδείας, της εκπαίδευσης και της καταχώρησης των γεννήσεων. Μια, πιο, μια μητέρα που έχει λάβει μεγαλύτερη παιδεία, μεγαλύτερη εκπαίδευση, έχει πιο πολλές πιθανότητες να προβεί σε καταχώρηση της γέννησης. Υπάρχει λοιπόν σαφώς μια σύνδεση. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Δεν θεωρείται δηλαδή θέμα διακριτικής μεταχείρισης αυτό οι γονείς έχουν τις ίδιες πιθανότητες να καταχωρήσουν ένα αγόρι όπως και ένα κορίτσι. Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εθνοτική προέλευση. Βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες όπου υπάρχουν αυτόχθονες πληθυσμοί, μειονότητες, αυτός ο κόσμος που είναι συχνά που δεν καταχωρίζει τις γεννήσεις των παιδιών τους. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουν την ίση, ίση αντιμετώπιση και τα παιδιά αυτά όπως και τα άλλα παιδιά τη εκάστοτε χώρας και να μην γίνεται αντικριτική μεταχείριση των παιδιών αυτών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι προφανώς ε, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με το εισόδημα. Όσο πιο υψηλό είναι το μισθολογικό επίπεδο των ατόμων, τόσο πιο ε, μεγάλες οι πιθανότητες Η πιο πλούσιοι <coughs> δηλώνουν τα παιδιά τους. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει ένα παιδί σε ηλικία, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να έχει δηλωθεί η γέννηση του. Όσο λοιπόν πιο δημοκρατική είναι μια κυβέρνηση και όσο πιο δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες για την εκλογή κυβέρνησης, τόσο πιο πολύ είναι εκεί το θέμα της ληξαρχικής πράξης γέννησης. Όσο λοιπόν εκδημοκρατίζεται μια χώρα και εκδημοκρατίζεται και η διαδικασία εκλογής ε, κυβέρνησης, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες. Είναι κρίμα όμως να περιμένει κάποιος μέχρι το 18 του για να αποκτήσει μια ταυτότητα, για να πιστοποιηθεί ότι υπάρχει καν. Και αυτό σε πολλέ περιπτώσει σημαίνει ότι το άτομο αυτό δεν έχει πρόσβαση σε ασφάλεια υγειονομική, σε κοινωνικές υπηρεσίες και το καθεξής. Τώρα, ποιε είναι οι μελλοντικέ προοπτικές. Θα δείτε εδώ πέρα ότι η χώρα η οποία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, οι χώρε μάλλον, είναι βασικά οι χώρε τη Ασία. Παγκλατές, ως επιτοπλίστων και αυτό χάρη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 1994 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UNICEF ξεκίνησαν το πρώτο πρόγραμμα καταχώρησης γεννήσεων στον κόσμο. Στη χώρα λοιπόν αυτή το Μπαγκλαντές ε, καταχώρησε λιγότερο από το 15% των γεννήσεων. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 51%. Το Πακιστάν, η Ινδία προφανώς με εξαιρετική πυκνότητα πληθυσμών έχουν σημαντικά προβλήματα. Στην Αφρική δε ε, Νιγηρία και Γκάνα, χώρες με γαλλόφωνη παράδοση, είχαν ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε. Θα πρέπει όμως να υποστηρίξουμε τις εθνικές κυβερνήσεις για να εξυγχρονίσουν και να θέσουν εκ νέου σε λειτουργία το σύστημα αυτό. Στην ε, Ανατολική και Νότια Αφρική το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα. Υπάρχει μια τεράστια ορμή σήμερα σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά τις καταχωρήσεις των γεννήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα σχετικά μη πολιτικό. Όλες οι κυβερνήσεις είναι πεπισμένες για τα ωφέλη. Έχουν ληφθεί λοιπόν πολλές πρωτοβουλίες από περιφερειακές οργανώσεις επίπεδο ΙΕ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα θα ζητήσω και από τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ που ξεκίνησε μια εταιρική σχέση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα έτος για να υποστηριχθούν κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες και στην Αφρική αλλά και στον Ελληνικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να ενθαρρυνθούν οι ευρωβουλευτές αλλά και οι βουλευτές της χώρας, της, της ε, εκάστοτε να προωθήσουν νομοθεσία και νομοθετικά πλαίσια προκειμένου να είναι δωρεάν, καθολική και έγκυρη η καταχώρηση των γεννήσεων. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Να εκχωρούνται πόροι για την καταχώρηση των γεννήσεων. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η καταχώρηση γεννήσεων θα ενταχθεί σε διάφορα άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάρενς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πίτερς γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας έκανε. Θα να μιλούμε για θεαματική πρόοδο σε θέματα καταχώρησης των γεννήσεων είναι σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε ορισμένε καταχρήσεις που γίνονται κατά την καταχώρηση των ε, νεογέννητων. Έχετε επίγνωση και έχετε αναλάβει μέτρα για το γεγονός ότι μερικές φορές ε, υπερβολική πληροφόρηση μπορεί να δώσει, υπερβολικό αριθμό πληροφοριών μπορεί να δημιουργήσει καταχρήσεις. Το είδαμε στη Ρουάντα που αναφέρονται και η εθνοτική προέλευση. Όταν γίνεται μια δολοφονία από το κράτο, όλες, ε, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, για να καταλήξουμε σε γενοκτονία κάνετε κάποιες προσπάθειες ώστε να μην αναφέρετε η εθνοτική ή η θρησκευτική προέλευση στις, ε, στις ταυτότητες ε, σε αυτές τις χώρες. Το έχετε σκεφτεί. Ευχαριστώ. Το, λόγο... το λόγο έχει η κυρία Μαρίνα Μαρκέτη από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζεται με την UNICEF στη προσήλωσή της στην προστασία των ε, δικαιωμάτων του παιδιού ε, παγκοσμίω και πρόκειται για την ε, πρώτη ενέργεια για την προστασία του παιδιού, η καταχώρησή του δηλαδή κατά τη γέννηση. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τη UNICEF σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο μόλις ανέφερε η Λίλα Ιδρύσαμε αυτό το πρόγραμμα σε 8 χώρες, Μπουργκίνα Φάσο, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Μιανμάρ και τρεις, χω... τρεις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, Βανουάτου, νησιά Σολομόντα και Κυριμπάτη. Στόχος είναι να αυξηθεί η καταχώρηση των γεννήσεων στις χώρες αυτές κατά τουλάχιστον 20% και να μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην καταχώρηση στις αστικές ε, και στις ε, γεωργικές περιοχές τουλάχιστον κατά 50%. Έχουμε λάβει την πρώτη ενδιάμεση έκθεση που ήδη μας δίνει πολύ θετικά αποτελέσματα, πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έχουν εκπαιδεύσει τις χώρες για το πώς να διαχειριστούν ε, το Μητρό και τα συστήματα στατιστικής, όπως στην Μπουρκίνα Φάζο μόλις δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα 30 νέων στατιστικολόγων, όπου εμείς παρέχουμε ε, την βοήθεια για την ε, συλλογή και διαχείριση των στοιχείων. Επίσης, στρατηγική για πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές έχει σχεδιαστεί με κινητές ταξιαρχίες που θα μεταβαίνουν και θα αναζητούν τα νεογέννητα που πρέπει να καταχωρηθούν, ιδιαίτερα για τη Μοζαμπίκη γι' αυτό που η UNICEF έχει καταγράψει πρόσφατα 740.000 παιδιά κάτω των 5 ετών που δεν είχαν ακόμα καταχωρηθεί. Στο Κιλιμπάτι, σε ένα μόλις χρόνο δραστηριότητα, οι ε, καταχωρημένες γεννήσεις αυξήθηκαν από το 68% στο 82%. Μόλις ένα χρόνο μετά, λοιπόν, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και πραγματικά βασιζόμαστε σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε μάλλον... Ε, βέβαια θα έχουμε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα σε άλλον ένα χρόνο. Συμμετέχουμε επίσης σε συζητήσεις για άλλους, άλλες πηγές για την καταχώρηση των γεννήσεων, όπως είπε και η Λίλα, ιδιαίτερα τα υγειονομικά συστήματα. Συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τελευταία εκ των οποίων διοργανώθηκε τον περσίνο Δεκέμβριο όπου συζητήθηκαν και πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα υγείας ώστε να ε, καταχωρείται το νεογέννητο. Διάφοροι πυρογνώμενες πρότειναν διάφορες δυνατότητες και η πιο θετική είναι η καταγραφή με το κινητό που βέβαια σημαίνει διάφορα προβλήματα γιατί έχουμε θέματα προστασίας των δεδομένων, έχουμε θέματα λογισμικού, τεχνικά, αλλά και προβλήματα αγραμματοσύνης. Γιατί πώς μπορεί ένας αγράμματος άνθρωπος να στείλει μήνυμα ότι πρέπει να κατακορυθεί το, τον του. Έχουμε λοιπόν διάφορα προβλήματα, θα πρέπει να γίνουν πιλωτικά προγράμματα και μετά ευρύτερα προγράμματα, αλλά εργαζόμαστε από αυτού. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε και τις παραδοσιακές γιορτές για την ονομασία του νεογέννητου θέλουμε για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τα νεογέννητα. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες λοιπόν. Συνεργασία με τη UNICEF θα γίνουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες με, υπό την ατζέντα για την αλλαγή που εστιάζουν στη σωστή διακυβέρνηση και φυσικά η προστασία του παιδιού και η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού θα είναι ένας βασικός άξονας της. Ευχαριστώ. Grazie Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο και πάλι στην κυρία Λίλα Πίτρη. σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Γκέρας για την ερώτησή σας. Και εγώ ήμουν στη Ρουάντα και πριν και μετά την γενοκτονία και σας διαβεβαιώ ότι μάθαμε το μάθημά μας από το πάθημα αυτό και σε όλες τις σχέσεις που έχουμε με όλες τις χώρες ε, όπου και βρίσκονται στον κόσμο προσπαθούμε να αποφύγουμε ε, να καταγράφεται τέτοια προέλευση εθνοτική ή να, αναφέρονται, ή να αναφέρεται η να η να αναφερεται η καταγωγη των αγωνιών και μάλιστα ε, δεν θέλουμε να αναφέρεται η στου προταστερατορισμός των γονιών, να απορρίπτεται η καταχώρηση σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί εκτός γάμου και το καθεξής. Σε όλες ε, τις σχέσεις μας με κυβερνήσεις και χώρες, αλλά και με τους περιφερειακούς φορείς, έχουμε δημιουργήσει ένα μορφότυπο, στερεότυπο για τις καταχωρήσεις των γεννήσεων. Στην περίπτωση του Βιετνάμ, για παράδειγμα, ή στην περίπτωση του Μπαγκλαντές, εκεί έχουμε αυτόχθονες κοινότητες που αρνούνται να καταχωρήσουν τα νεογέννητά τους εξαιτίας αυτής της ύπαρξης. Αλλά το θέτουμε συνέχεια στο διάλογο το θέμα αυτό. Και μέχρι στιγμής και από το 2005 όταν βλέπω τα νέα έντυπα για την καταχώρηση των γεννήσεων βλέπω ότι πραγματικά έχουμε επιτελέσει θεαματική πρόοδο. Φυσικά η πρόκληση είναι να υιοθετήσουν οι κυβερνήσει το νέο σύστημα, όπω ανέφερε και η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή. Αυτή είναι η σημαντική πρόκληση. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Δεν αναφερθήκατε στην θρησκεία. Το θρήσκευμα τελικά αναφέρεται. Ναι, ούτε το θρήσκευμα αναφέρεται. Στην περίπτωση αυτή, στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, που έχουμε και χριστιανούς, ε, εβραίους ε, και μουσουλμάνους, για τους ενήλικες υπάρχει σημαντικό εδώ θέμα. Θα σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην Ορδανία προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στου γονείς, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί λένε στη δική μου ληξιαρχική πράξη γέννηση αναφέρει το θρήσκευμα. Γιατί στην ληξιαρχική πράξη γέννηση του παιδιού μου να μην αναφέρεται. Προσπαθούμε πάντω να ευαισθητοποιήσουμε και του κρατικού φορεί, αλλά κυρίω του γονεί. γιατί επιμένουμε στην αρχή του δικαίου, ότι θα πρέπει να υφίσταται διακριτική μεταχείριση ένα παιδί ή να καταβαλτούνται οι αρχές δικαίου. Να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκεύματος και το καθεξής. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στα σημεία 14 και 15 που προτείνω να τα εξετάσουμε από κοινό. Αυτά αφορούν τη γνωμοδοτής της Επιτροπής μας για την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Επιτροπή, για την εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού της Ένωσης και για την ε, εφαρμογή εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για το 2012. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι βεβαίως η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού που ξεκίνησε την εργασία του μετά από την δημοσίευση της έκθεσης των ετησίων μάλλον εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Νοέμβριο. Στη δική μας Επιτροπή αυτές οι γνωμοδοτήσεις παραδοσιακώς προετοιμάζονται από τον ίδιο βουλευτή που υπήρξε και εισηγητής για την απαλλαγή απαλλαγή ε, μάλλον γιατί το έτος αυτό, το 2012. Και το 2012 υπεύθυνος ήταν ο κύριος Γκέρενς και θα του δώσουμε αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως προτείνατε, θα παρουσιάσω και τις διεκθέσεις την έκθεση για την απαλλαγή για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αυτό που είναι σημαντικό για την απαλλαγή, για να το πούμε απλά, αν δεν βρούμε κανένα με το χέρι στη τσέπη, με το χέρι στο ταμείο και από τους δωρητές και από τους αποδέκτες, θεωρούμε ότι ήδη είναι κατά το ίμιση επιτυχής η δράση, αν δεν πιάσουμε κάποιον στα πράσα δηλαδή. Και ε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την αναπτυξιακή δράση. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των σφαλμάτων και των συγκεκριμένων περιστατικών. Ε, φυσικά και τα σφάλματα δεν είναι αμεληταία, γιατί ένα σφάλμα μπορεί να είναι συστημικό, να έχει συστημικό χαρακτήρα σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Γιατί κάθε σφάλμα που έχει αποκαλυφθεί και που έχει αποτελέσει το... έχει γίνει είδηση, ουσιαστικά κυλιδώνει όλη την αναπτυξιακή συνεργασία και όλες τις ε, σχετικές δράσεις. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα οξυδερκείς και να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγουμε τα λάθη. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είμαστε και υποκριτές. Θα πρέπει να γίνει διάκριση λοιπόν μεταξύ συστηματικής διαφθοράς, ληστρικής διαφθοράς, αρπακτικής των λεγόμενων ελίτ που βάζουν χέρι σε πλούτο που δεν τους ανήκει. Και να κάνουμε το διαχωρισμό από αυτή τη συστηματική, συστηματική διαφθορά και την ε, μικρή σεβέλη διαφθορά κάποιου υπαλλήλου που προσπαθεί να συμπληρώσει κάπως ε, το πενιχρό εισόδημά του. Και στην αναπτυξιακή βοήθεια έχουμε συνήθως ε, τέτοιου είδους μικροδιαφθορά να αντιμετωπίσουμε. Η Όλαφ έχει αναλύσει 45 περιπτώσεις, έχει γίνει καταγγελία σε 45 περιπτώσεις στην Όλαφ, ε, με θέμα και την διπλή χρηματοδότηση. Και εδώ έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει περίπτωση διπλής χρηματοδότησης σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο και ταυτόχρονα συγχρηματοδοτείται αυτό από συγκεκριμένο κράτο. Αν δεν έγινε ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτου μέλου, ίσω ε, δημιουργηθεί τέτοια επικάλυψη, γιατί είχαμε τέτοια διπλή χρηματοδότηση στο παρελθόν. Υπάρχει τώρα ένα σύστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον για να αποφευθούν τέτοιου είδου ε, διπλές χρηματοδοτήσει. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει μία σωστή κατάρτιση καταλόγου χρηματοδοτήσεων για να αποφευθούν τέτοιες διπλές χρηματοδοτήσεις γιατί όταν λαμβάνουν χώρα πραγματικά πλήττουν την αξιοπιστία της αναπτυξιακής πολιτικής. Και μετά μιλούμε και για το RER, το εναπομείναν ποσοστό σφάλματος. Αυτό το εναπομείναν ποσοστό σφάλματος αφορά λάθη που δεν αποκαλύφθηκαν, δεν επισημάνθηκαν. Βέβαια αυτό το ΡΕΡ μειώνεται σημαντικά. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γενικό προϋπολογισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Έχω την ίδια πορεία που είχα και για το γενικό προϋπολογισμό η Όλαφ μπορεί να επιληφθεί περίπτωση που αφορά το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Γιατί το ΕΤΑ δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι, ανήκει στα κράτη-μέλη και στην ΑΚΕ, στην Ισομπερή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι εκτελεστικός φορέας ουσιαστικά και έχει εντολή από τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείρισή της και εδώ κάνω παρατήρηση και όχι ερώτηση πιστεύω ότι έλαβε υπόψη τις συστάσεις που κάναμε και τα σχόλια επίσης του ελεκτικού συνεδρίου. Φαίνεται ότι η δημοσιονομική ενίσχυση αφορά το 30% του συνόλου των κονδυλίων, κάτι που συνιστά σημαντική πρόοδο. Έχει αυξηθεί κατά 90% και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον έλεγχο στις χώρες που δέχονται τέτοια, λαμβάνουν τέτοια δημοσιονομική υποστήριξη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δούμε πώς λειτουργεί εμπράκτος αυτός ο έλεγχος και που έγκυται η πρόοδος. Και εδώ όμω ε, έχουμε κάποια λάθη που παρόλα αυτά έχουν μειωθεί από 5,1 σε 3% το ποσοστό εναπομείναντος σφάλματος σε σχέση με τα συνολικά κονδύλια που έχουν καταβληθεί. Πάντως αναφέρω στο ψήφισμα ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συγκεκριμενοποίηση της θέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου με τον έλεγχο που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ε, μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Περιμένω λοιπόν την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την ευθυγράμμιση. Αυτή είναι μια παλιά απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το να ενταχθεί το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω. Κάθε φορά μας υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μέχρι το 2020 θα υποβληθεί μια λύση, αλλά δεν ξέρω σε τι φάση βρισκόμαστε προ προς την εκπόνηση αυτής της λύσης. Πολύ φοβάμαι ότι ο ορισμός που έδωσε ο Δεκόλ για τον ορίζοντα Ίσως ε, ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Ο Ντεγκόλ είπε ότι ο ορίζοντας είναι μια γραμμή που υποχωρεί στο μέτρο που εμείς προχωρούμε. Και πολύ φοβούμαι ότι η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών ε, ως προς τον ορίζοντα του πότε θα υποβληθεί η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται δυστυχώς στον ορισμό που έδωσε ο Ντεγκόλ για το TST ορίζον. Σας ευχαριστώ πολύ για την αδιάλειπτη προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο ο κύριος Μισελ. Μίτσελ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να το πω και να μην με παρεξηγήσετε, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό στην αναπτυξιακή βοήθεια να προσπαθούμε να έχουμε αποτελεσματικότητα, οικονομία και αποδοτικότητα. Όμως, δεν μπορούν όλα να πηγαίνουν σωστά και όλα να είναι τέλεια. Γιατί ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να γίνεται με βάση εμπιστοσύνη και αμεσότητα και αν υπήρχε ένα πρόβλημα, μάλλον αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα στην οικονομία και την αποδοτικότητα και το να ταΐσουμε τον κόσμο, εγώ λέω να ταΐσουμε τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ένας βαθμός αβεβαιότητας σε αυτό το προϋπολογισμό πάντα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ελαστικότητα στους κανόνες της προσπάθειας ελέγχου των δαπανών γιατί, ε, και των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν πού πήγαν τα χρήματά τους. Αυτό είναι πρώτο και κύριο επίσης. Όμως ε, πρέπει να σκεφτούμε όσο γίνεται με βάση αυτά τα τρία που είναι τα χρηματα οικονομία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Οικονομία τι σημαίνει, ποιο είναι το πιο φθηνό ε, φάρμακο που να είναι όμως και ποιοτικό. Γιατί εντάξει μπορεί να βρεις κάτι πολύ φθηνό αλλά μην είναι ποιοτικό. Αλλά αν επιμείνουμε στην ποιότητα, ποια είναι η καλύτερη τιμή που μπορούμε να έχουμε. Από, αποτελεσματικότητα, ας πούμε, αν ένα μπουκάλι ε, ε, εμβολίου φτάνει για 20 εμβόλια, να δούμε αν όντω κάναμε 20 εμβόλια και επί αποθετικότητα είναι μειώσαμε τα περιστατικά της τάδε ασθένειας, ας πούμε πολιομελίτιδα ή οτιδήποτε, με βάση το στόχο που είχαμε θέσει πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν να το σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε περισσότερο με αυτόν τον τρόπο καθώς προχωρά ο καιρός και έπειτα να πούμε και ότι είναι και τμήμα της ανθρώπινης φύσης ότι όταν ε, κυκλοφορεί πολύ χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, όταν ε, πολύ χρήμα κυκλοφορεί λοιπόν ε, και είναι η ανθρώπινη φύση λοιπόν να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι περνάει το... εμείς θα πρέπει αυτό να το αναμένουμε και να το εμποδίσουμε αν μπορούμε και να φροντίσουμε ε, γιατί εδώ υπάρχουν ε, ενδείξεις ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί. Ο εισηγητής μιλάει για την αξιολόγηση, τον αντίκτυπο και την παρακολούθηση και πώς αυτά γίνονται με βάση την οικονομική διαχείριση είναι σημαντικό και θέλω να το στηρίξω. Ε, επίσης καλωσορίζομαι το γεγονός ότι υπήρχε μείωση στον αριθμό των προγραμμάτων, μείωση του αριθμού των προγραμμάτων που είχαν μεγάλα προβλήματα από το 8% το 2010 στο 5% το 2012. Αυτή είναι σημαντική μείωση και καλό σημάδι. Καταλαβαίνω ότι ο Ιναπών του όσον αφορά το αναπτυξιακό ταμείο. Κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε έναν ε, υπάλληλο σύνδεση, έναν αξιωματούχο σύνδεση, κάτι εν πάση περιπτώσει, ώστε να συνεργαστούμε με πιο συγκεκριμένο δομημένο τρόπο και να πιέσουμε το Συμβούλιο. Είναι σκανδαλώδε ότι δεν μπορούμε πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια μέσω τη στενότερη συνεργασία. Ε, Αφού δεν χρειάζεται να τα αναλάβει όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να αναλάβει η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Βρετανία ή η Κομισιόν αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε τις εμπειρίες μας. Γιατί βλέπουμε ότι 800 εκατομμύρια ευρώ χάνονται στα κόστη συναλλαγών λόγω τη επικάλυψης που υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας γιατί είναι πραγματικά απογοητευτικό που το ε, Αναπτυξιακό Ταμείο μένει εκτός του δικού μας ελέγχου. Καλωσορίζω τις μεταρρυθμίσεις και τη σταθερότητα στο κέρας Αφρικής και την ε, Βραζιλία και, και την μείωση του κινδύνου καταστροφών. Όταν μιλήσαμε για αυτά τα, την αποτελεσματικότητα, την οικονομία και την αποδοτικότητα, αν κανείς δαπανίσει για την ε, φυσική, να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές, από τη στιγμή που χτυπά μια τέτοια φυσική καταστροφή, το κόστος μπορεί να είναι τεράστιο. Από ανθρώπινη πλευρά, από οικονομική πλευρά, από φυσική καταστροφή. Και έχει ε, ε, για κάθε ευρώ που δαπανάτε για τη μείωση ε, του κινδύνου της καταστροφής ε, αποδίδει 4 ευρώ ε, και στη δική μου έκθεση σημαίνει ας πούμε ότι χτίζουμε και σχολεία σε πιο ασφαλή μέρη κτλ. Στη Κίνα φάνηκε ένα, εκατομμύριο, ένα ευρώ αποδίδει 4 εκατομμύρια. 12 δις λέει εξοικονόμησαν στην Κίνα η Κομισιόν αυτό το προωθεί. Και νομίζω πως για το νέο κοινοβούλιο η μείωση κινδύνου ε, σε περίπτωση καταστροφής και η αντοχή και η δαπάνη των αναπτυξιακών χρημάτων για τέτοιους σκοπούς θα πρέπει να είναι ε, πολύ σημαντικότερη. Σας ευχαριστώ. Grazie, σας ευχαριστώ. Σας, ε, και τώρα δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή του κύριο Λουκ Μπαγκμπούρ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκέρενς για τις γνωμοδοτήσεις του σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού για τις απαλλαγές στο Γενικό Προϋπολογισμό και στο ΕΤΑ, το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Και μάλιστα τονίζονται και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό σφάλματος που διαπιστώθηκε στον προϋπολογισμό, μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του ποσοστού σφάλματο που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο οφείλεται στην αλλαγή τη μεθοδολογία. Αν δεν είχαμε αλλάξει τη μεθοδολογία, το ποσοστό σφάλματο θα ήταν κάτω του 1%. Θεωρούμε ότι ο τρόπος υπολογισμού του εναπομείνοντος ποσοστού σφάλματος ε, που έχει θετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χρήσιμος ε, αυτός ο υπολογισμός, ε, η μέθοδος υπολογισμού και χαίρομαι που και το ελεκτικό συνέδριο αναγνώρισε τη, τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθοδολογίας. Με την έκθεση αυτή εντοπίσαμε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και Υιοθετήσαμε και ένα σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε πέρυσι την Άνοιξη και που θα μας επιτρέψει να διορθώσουμε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Και λάθη, κυρίως λάθη που έγιναν σε πληρωμές σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά το ΕΤΑ, παρόλο που το ποσοστό σφάλματος είναι άνω του 2%, υπάρχει μια μείωση από 5% στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτό το ποσοστό κάτω από 2% ή γύρω στα 2%. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Γκέρενς ως προς την ΟΛΑΦ και η σχέση ΟΛΑΦ και ΤΑ, Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η ΟΛΑΦ έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες είναι σε θέση να διαβιβάσουν την ΟΛΑΦ κάποιες υποθέσεις για να τις εξετάσει. Και μάλιστα έχουμε αύξηση των περιπτώσεων αυτών, γιατί οι υπηρεσίε είναι όλο και πιο ευαίσθητε. Και όταν υπάρχει υπόνοια για μία συναλλαγή, για μία δράση, προτιμούμε να ε, παραπέμπουμε το θέμα στην Όλαφ για να έχουμε μία σαφή απάντηση για την ε, νομοτυπία και την ορθότητα των συγκεκριμένων δράσεων και πληρωμών. Σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο, η πρόταση αυτή έγινε στην ανακοίνωσή του σας και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έγινε δηλαδή μια πρόταση να ευθυγραμμιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας με τον έλεγχο για το ΦΕΔ, για το ΕΤΑ. Θα ληφθεί απόψε στις ε, προτάσεις που θα κάνουμε για τις ε, προτάσεις αναπτυξιακής βοήθειας. Και τώρα η συμπερίληψη του ΦΕΔ στον προπολογισμό εξακολουθεί να είναι στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έχουμε διατρανώσει. Και μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχαμε προτείνει για πρώτη φορά την ένταξη του ΕΤΑ στον προπολογισμό. Και έκτοτε συστηματικά προτείνουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς ε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι στην περίοδο μετά του Κοτονού και μετά το 2020, πριν από το 2020 που θα ολοκληρωθεί και το 10ο έτα, να έχουμε εξέλιξεις. Σε ό,τι αφορά την διπλή χρηματοδότηση. Και αυτό το θέμα μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό με διάφορα εργαλεία που έχουμε και μηχανισμούς. Καταρχήν ο συντονισμός επιτόπου μας επιτρέπει να αποφύγουμε διπλή χρηματοδότηση με διάλογο και συνεργασία. Επίσης υποβάλλουμε στα κράτη-μέλη ε, τα προγράμματα σε πρόωρο στάδιο και υπάρχει φυσικά έλεγχος και εξάντε και εξ που γίνεται επί τόπου. Έτσι εντοπίζουμε τις περιπτώσεις διπλής χρηματοδότησης. Πάντως, τέτοιες περιπτώσεις διπλής χρηματοδότησης σήμερα τουλάχιστον είναι σπάνιες. Τώρα, για κάποιες ε, ε, για τη συζήτηση που είχαμε για τη δημοσιονομική υποστήριξη. Έγιναν σφοδρές συζητήσεις ε, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελικά είχαμε μια ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική υποστήριξη μετά από έντονε συζήτηση και στο Συμβούλιο και μετά από το ψήφισμα το σχετικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα νέα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε την θέση της και θέσπισε νέα εργαλεία, πολύ καλύτερα προσαρμοσμένα στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια και στο μηχανισμό αυτό της δημοσιονομικής υποστήριξης. Έχουμε για παράδειγμα συμβάσεις ε, για την ανασυγκρότηση του κράτους δικαίου ή για την ανασυγκρότηση του κράτους ε, σε περίπτωση ευπάθειας. Έχουμε μεγαλύτερο σύνδεσμο με τα θεμελιώδη δικαιώματα και γίνεται ενδελεχής ανάλυση εκ των προτέρων της κατάστασης του εταίρου μας για να ληφθεί απόφαση για το κατά πόσο θα δοθεί αυτή η δημοσιονομική στήριξη. Επίσης γίνεται καλύτερη ανάλυση των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη και τη στάση του ελεκτικού συνεδρίου και των αντίστοιχων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι στιγμής είχαμε 73 ε, μελέτες για τα χαρακτηριστικά κινδύνου που μπορεί να έχουν οι εταίροι μας, το προφίλ κινδύνου και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα και αυτά τα σημεία έχουν ενισχυθεί. Και δεν έχουμε μόνο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που είναι σημαντικός γιατί θέλουμε ε, η πολιτική και ο προϋπολογισμός να συζητώνται και να εγκρίνονται από ε, όργανα που χαρακτηρίζονται από εκπροσώπηση και στις ε, χώρες εταίρους, αλλά τονίζουμε και την ε, ανάγκη εξωτερικού ελέγχου από το ελεκτικό συνέδριο ή από ανεξάρτητους ελεκτές, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνεται σωστή χρήση των κονδυλίων της κυβερνήσης. Ό,τι αφορά την αλυσίδα της διαχείρισης των δημόσιων λογαριασμών, από την θέσπιση του προϋπολογισμού μέχρι την εκτέλεσή του και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων. Να εξασφαλίσουμε έλεγχο σε όλα τα στάδια. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Κέρενς για να κλείσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή αλλά και τον συνάδελφο Γκέι Μίτσελ για τα σχόλιά του. Νομίζω πως συμφωνούμε επί τη ουσία. Ο Γκέι Μίτσελ λέει πω υπάρχουν δύο διαστάσεις λογιστική και η πολιτική. Θα τη λάβουμε υπόψη. Θα έλεγα ότι και όσον αφορά την απαλλαγή, ποτέ δεν υπάρχει μηδενικό κίνδυνο όσον αφορά την πολιτική αναπτυξία και συνεργασία. Αντίθετα, η αποκάλυψη ενός λάθους επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου. Εάν δεν βρούμε κανένα λάθος, εγώ ανησυχώ περισσότερο από το αν αποκαλυφθεί ένα σφάλμα και πρέπει να έχουμε και την αίσθηση των διαστάσεων και των όγκου καθώς και των λίγων ανθρώπων που ασχολούνται με την εκτέλεση των πολιτικών και όπου τα σφάλματα είναι εξαιρετικά λιγοστά από αριθμητική άποψη. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. λιγότερο στην Κομισιόν επικρίνω από ότι εμάς τους ιδίους είμαστε άχρηστοι. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει με τα Εθνικά Κοινοβούλια να φτιάξουμε ένα σύστημα ελέγχου του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Ανάπτυξης και τα κράτη άχρηστα τα Εθνικά Κοινοβούλια μάλλον άχρηστα, γιατί κανένα μέχρι τώρα δεν κάλεσε τον αρμόδιο επίτροπο να λογοδοτήσει ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου του. Ε, ενώ είναι κοινή ε, ιδιοκτησία όλων των κρατών μελών το Ταμείο αυτό και τα άρα τα κράτη-μέλη έχουν απόλυτα το δικαίωμα να καλέσουν τον Επίτροπο και μάλιστα το είπα και στον Πιπάρξ και μου το επιβεβαίωσε και αυτός. Προσπάθησα να πειράξω κάπως ε, και το κοινοβούλιο της χώρας μου που είπαν «Ε, ναι, ναι θα το κάνουμε, το μεταξύ έχουμε νέα πλειοψηφία οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και πάλι. Εμείς πρέπει λοιπόν να συνοηθούμε για έναν αξιωματικό σύνδεση, σε πάση περιπτώσει, ας είμαστε φάνταστοι και αποτελεσματικοί, δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει και να συνεννοηθούμε για ένα σύνολο στόχων, για θέματα, αλλά και για κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να πάψει αυτή η γνωστή αυτή αναποτελεσματικότητα. Επιμένω τώρα όσον αφορά τη διπλή χρηματοδότηση. Εδώ το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχει σε επίπεδο της Κομισιόν ένας πλήρης κατάλογος όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται από τα κράτη-μέλη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι θα ήταν το λιγότερο αυτό. Κάθε κράτος μάλλον να κοινοποιεί στην Κομισιόν το σύνολο των προγραμμάτων του, όσα προγραμματίζει, όσα είναι υπό εκτέλεση, ώστε να έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να συγκρίνει τη δράση της με αυτή των κρατών μελών για να δούμε πως υπάρχει επικάλυψη και συγχρηματοδότηση. Ο διάλογος των ε, χωρών ε, αποδεκτών είναι καλός, αλλά δεν αρκεί. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου τώρα να σας θυμίσω πως η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για αυτά τα δύο σχέδια γνωμοδότησης είναι η 5η 23 Ιανουαρίου στις 18 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου επόμενο μας σημείο είναι και κλεισμένο το θυρών. Μόνο βουλευτές λοιπόν, η βοηθή του, συνδιαπιστευμένοι, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, καθώς και το προσωπικό της γραμματείας μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα. Θα ζητήσω λοιπόν από όλους τους άλλους να εξέλθουν τις αιθούσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. L'incontro Η δημόσια συνεδρία θα συνεχιστεί το απόγευμα στις 3 στην ίδια αίθουσα.